So, Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, ξεκινάμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε σήμερα ένα μεγάλο εκτενές πρόγραμμα και θα ήθελα από κοινού να το πάρουμε, να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε αν συμφωνείτε. Έγκριση ημερήσιας διάταξης και μετά εξή πληροφορία ανακοινώσεις Προέδρου. Το σημείο 15, Μωρέ Σαντιέ, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα το εξετάσουμε μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Αμέσως μετά θα έχουμε την ημερήσια διάταξη που θα ξεκινήσει και θα συνεχίσει κανονικά. Μετά έχουμε το σημείο 6 του συναδέφου μας Μπουλόν ε, σχέδιο γνωμοδότησης για την εκβιομηχάνηση, νέα εκβιομηχάνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το εξετάσουμε και αυτό. Αλλά μετά το 12, μετά το 12 και για το σημείο 7 είναι η έκθεση Προέδρου μας της κυρίας Μπερές σε σχέση με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και στον έλεγχο των κρατών μελών για την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Για να συνειδητοποιήσει κανείς τι σημαίνει σε μετάφραση αυτός ο τίτλος. Αυτό αφαιρείται, αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη. <clears throat> Θα ψηφίσουμε μένα, αλλά δεν θα εξετάσουμε τώρα τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε. Έχει ληφθεί αυτή η απόφαση, είναι σαφής. Ελπίζω ότι συμφωνείτε. Εξέταση τροπολογιών λοιπόν για την έκθεση αυτή λέει σύμφωνα με το 81 θα προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη αύριο πριν από το σημείο 14. Αύριο πριν από το 14. Η τελευταία πληροφορία που μπορώ να σας δώσω σχετικά. Εγκρίθηκε λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Έτσι μπορούμε να το πούμε αυτό. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Επόμενο σημείο σύντομα να σας αναφέρω ανακοινώσεις Προέδρου πολύ γοργά για την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη μια κοινή συνεδρίαση μεταξύ δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών της Απασχόλησης και της ΕΚΟΝ. Στο Στρασβούργο στις 21 Νοεμβρίου θα έχουμε μια έκτακτη ξεχωριστή συνεδρίαση από τις 8 και 4 έως τις 10 ο Επίτροπος Ρεν και ο Επίτροπος Άντορ και οι δύο Επίτροποι από κοινού θα παρουσιάσουν την ετήσια αυτή έκθεση για την ανάπτυξη που από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάστηκε από, την 13, ε, τις 13 Νοεμβρίου θα έχει εξαρταστεί και καλυφθεί. Είναι σημαντικό αυτή την ημερομηνία τη σημειώσετε στα, στις ατζέντες σας, στα ημερολόγια σας ε, για το, την ε, διερμηνία, για τη μετάφραση. Είναι σημαντικό και η χρήση όσον αφορά τη διαδικασία ε, συμφιλίωσης, συμ, συνδιαλλαγής. Μου φαίνεται ότι λειτουργικά πάνε τα πράγματα, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση και αυτό είναι επίση σημαντικό. Οι ευρωβουλευτέ αποσαφηνίζεται ότι κάνουν πάντα καλές εκθέσεις και καλές παρεμβάσεις πρέπει να κάνουν. Βρισκόμαστε στο διαδίκτυο. Το μισό τη υφηλίου παρακολουθεί τα όσα κάνουμε και τα τεκτενόμενα και τις παρατηρήσεις μας και για τους συναδέλφους θα ήθελα να πω σήμερα πιέζει ιδιαίτερα ο χρόνο. Για κάθε θέμα θα έχουμε μόνο 15 λεπτά συνολικά για κάθε θέμα τη ημερήσια διάταξη. Όντα σύντομοι μπορούμε να αποδείξουμε σήμερα και να καταδείξουμε στου πολίτε οι ευρωβουλευτές καμιά φορά πολύ γοργά μπορούν να ολοκληρώσουν σημεία τη ημερήσια διάταξη. Θα το κάνουμε αυτό σήμερα σίγουρα. Μετά το 3 έχουμε το 4. Η κυρία Ελιζαμπέτ Μογάν Σαντιέ έχει τον λόγο. Παρακαλώ έχει τον λόγο Ελιζαμπέτ. Ε, Ένα σημείο για το τελευταίο τριμερή διάλογο που είχαμε είναι ο 26ος. Θα υπάρξει και 27ος την επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα πολύ σύντομα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τους διοικητικούς μας υπαλλήλου και όλη τη διαπραγματευτική ομάδα που κρατάει τον πύχη ψηλά. Ε, επίσης δουλεύει άεργα. Ε, Εργοδό, συγγνώμη. Ε, ο τελευταίος τριμερής διάλογος τελείωσε μία μισή ώρα το βράδυ. Θέλω λοιπόν να τιμήσω όλους όσους συμμετείχαν, να τους ευχαριστήσω θερμά. Στην τελευταία μας, στο τελευταίο διάλογο, όλα τα σημεία συμφωνίας τα διατρέξαμε πολύ γρήγορα. Σας έχω μιλήσει για αυτά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αλλά ε, είδαμε ποια είναι τα δύσκολα σημεία που μας μένουν. Τώρα είμαστε στο πιο δύσκολο τμήμα της διαπραγμάτευσης και επί των σημείων αυτών έχουμε πάρει όλη θέση. Το πρώτο δύσκολο σημείο. Το 25% του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να πάει στο Κοινωνικό Ταμείο. Η διαπραγματευτική σας ομάδα και η συγκήτριά σε αυτό το σημείο δεν έχουν ε, εγκαταλείψει τις θέσεις τους και ξέρουμε ότι έχουμε μαζί μας την υποστήριξη του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών, του Αλέν Λαμασούρ, και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι πολύ ευνοϊκό στο αίτημά μας. Συνομίλησα και με τον πρόεδρο της πολιτικής μας ομάδας, με τον Τζόζεφ Ντόλ, Προσπαθούμε λοιπόν όλο το βάρος που μπορούμε να έχουμε σε αυτή τη μεγάλη διαπραγμάτευση, θέλουμε να το, να το, ασκήσουμε. Να το ασκήσουμε. 11 ε, δισεκατομμύρια ευρώ είναι το διακύβευμα για το ανθρώπινο δυναμικό. Δεύτερο σημείο. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Θα θυμάστε ότι στο κείμενο οι, δικαι... περιοχές που είναι δικαιούχοι είναι αυτές που έχουν πάνω από το 25% νέων ανέργων μεταξύ 15 και 25 χρονών. Θα θέλαμε να βάλουμε και περιοχές που έχουν πάνω επίσης από το 22,9% νέων ανέργων. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό Ξέρουμε βεβαίω ότι δεν πρέπει να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, όλα τα σημεία τη διαπραγμάτευση τα δικά μας να τα περάσουμε, αλλά θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί έχουμε και άλλα αιτήματα. Θυμάστε τις ε, τροπολογίες που έχουμε θέσει για αυτό το θέμα. Επέκταση μέχρι τα άτομα που έχουν φτάσει στο 30 χρόνο, στο 30 έτος ηλικίας τους. Ένα από τα δύο μπορούμε να τα περάσουμε. Τρίτο σημείο. Θα θέλαμε το Συμβούλιο να εγκαταλείψει τους δισταγμούς του και να πετύχουμε το 20% του κοινωνικού ταμείου, το οποίο θα πηγαίνει ε, για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και αυτό είναι πνεύμα της διαπραγματευτικής μας εντολής. Και τελευταίο σκληρό σημείο, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι πρόσφυγες να επανενταχθούν στους δικαιούχους του Κοινωνικού Ταμείου. Αυτά είναι τα σημεία διαπραγματευσής μας. Εκεί επικεντρώνουμε τις προσπαθίες μας με συντεταγμένο τρόπο. Δεύτερη πληροφορία. Θα θυμάστε ότι προσπαθούσαμε στο σχέδιο προπολογισμού του 2014 να περάσουμε την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ή όπου είχαν εγγραφεί οι πιστώσεις και στο σχέδιο προπολογισμού λοιπόν του 2014, 3 δισεκατομμύρια 400.000 ευρώ έχουν εγγραφεί στις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων και 2 εκατομμύρια 600.000 ε, θα πάνε για το 2015, τα υπόλοιπα δηλαδή. Μας περιμένουμε δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, τα προγράμματα, αυτά τα έργα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2014 και το 2005. Ο 27 ο τριμερής διάλογος θα γίνει την επόμενη Τρίτη. Και ελπίζουμε ότι θα τελειώσουμε πριν φτάσουμε στους 30 τριμερείς διαλόγους, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το ότι επιλέξαμε την Ελιζαμπέτη ήταν μια καλή απόφαση από πλευράς μας. Πραγματικά τα πράγματα είναι σε σίγουρα ασφαλή χέρια, εξαιρετικά. Υπάρχει κάποια πρόσθετη ερώτηση. Ο κύριος Θέρκας έχει τον λόγο. Παρακαλώ κύριε Θέρκας. Δεν είναι τόσο ερώτηση, αλλά κυρίως θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο έργο της διαπραγματευτικής ομάδας που έχουμε. Η Ελισαβέτ ξέρει ότι τη στηρίζω απόλυτα στηρίζω απόλυτα τη στρατηγική που ακολουθεί, την τακτική της. Απλώς, για να... Α, δεν το ξέρει μάλλον, να σας πω ότι σχετικά με τα δύο θέματα που μας απασχολούν κυρίως, προκειμένου να επεκταθεί η πρωτοβουλία για τους νέους, είτε σε περισσότερους νέους είτε σε περισσότερες περιφέρειες, γιατί δεν μπορεί να το κρατήσουμε περιορισμένο αυτό το πρόγραμμα. Αν πρέπει να επιλέξουμε επέκταση σε αριθμό νέων ή γεωγραφικά, εγώ θα έλεγα να το επεκτείνουμε στους νέους 27 με 30 ετών, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε ότι μια πρωτοβουλία για τους νέους αφήνει απ' έξω τους μισούς περίπου νέους που ψάχνουν δουλειά σήμερα και που είναι 27 με 30 ετών. Να ξέρεις λοιπόν ότι έχεις την πλήρη υποστήριξή μου, Λιζαβέτα. Ευχαριστώ θερμά. Άλλες ερωτήσεις, άλλες παρεμβάσεις. Παρακαλώ εσείς. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συνεχίσω ακριβώς σε αυτό που από πλευράς προλαλήσαντος ακούσαμε. Επέκταση αυτής της πρωτοβουλίας, διεύρυνση όσον αφορά τα άτομα μέχρι το 30ο του έτος ηλικίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελευταία ενέκρινε την έκθεσή μου και η έκθεσή μου ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να κινητοποιηθούν, αυτές οι προτάσεις να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν. Τον τελευταίο καιρό είχα και συνάντηση με τον Επίτροπο Άντορ πρόσφατα και έχω την εντύπωση ότι δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί ιδιαίτερα σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είναι υπέρ ώστε αυτή η πρωτοβουλία να επεκταθεί μέχρι το 30ο έτος ηλικίας. Ελίζαμπετ, η ερώτηση είναι προς εσένα. Υπάρχει ευκαιρία να υλοποιηθεί αυτό που πρότεινες. Μπορεί να εφαρμοστεί. Τι λες. Ευχαριστώ. Άλλη παρέμβαση, παρακαλώ. Δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση. Ωραία. Η Ελιζαμπέτ έχει τον λόγο να απαντήσει. Παρακαλώ, πολύ σημαντικά θέματα. Μπορεί να επεκταθεί μέχρι το 30ο έτος ή όχι. Τι λες. Ε, δύο λόγια μόνο. Πράγματι, συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα αυτή να επεκταθούμε ε, και να συμπεριλάβουμε και τους νέους που είναι μέχρι 30 ετών, γιατί πραγματικά δεν θα, θα ήθελα να αφήσουμε απ' έξω αυτήν την ηλικιακή κατηγορία. Η δυσκολία προέρχεται από τον αριθμό των νέων 25 με 30 που βρίσκονται στην ανεργία. Και αυτό για το οποίο με κατηγορούν στην πρόταση αυτή είναι ότι έτσι κινδυνεύουμε να αποδυναμώσουμε τις ε, επιπτώσεις, τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η πρωτοβουλία. Για να είμαστε λοιπόν αποτελεσματικοί, ζητάω καλό συντονισμό ανάμεσα στην πρωτοβουλία για τους νέους και την εγγύηση για τους νέους γιατί στοχεύουμε το ίδιο κοινό. Στην εγγύηση για τους νέους, να ξέρετε, έχουμε κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τις 101 περιοχές που έχουν άνεργους στην κατηγορία 15 με 25 και παραπάνω, αλλά αφορά το σύνολο των περιφερειών. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει καλή διάρθρωση μεταξύ των δύο. Εφόσον υπάρχει καλός συντονισμό με την εγγύηση για τους νέους, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Πάντως να ξέρετε ότι θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλες τις πολιτικές ομάδες για την συμπαράσταση που έδειξαν μετά από 26 τριμερούς διαλόγους, τριμερείς διαλόγους να ξέρετε ότι έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε καλά μεταξύ μας. Μάλιστα. Το να μπορεί κανείς να εργαστεί καλά με άλλα θεσμικά όργανα απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά, αλλά τα κατάφερες Ελίζαμπεθ. Ευχαριστούμε πολύ καλά και για την αλληλεγγύη που μπορέσαμε να έχουμε στην Επιτροπή μας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξη. Πρόκειται εδώ για την Σάρι Εσάγια, την εισηγήτρια Σάρι Εσάγια είναι η ταξινόμηση και επισήμανση για τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων. Έχει τον λόγο, Σάρη, για αυτέ τι τροπολογίε που έχουμε και το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε δύο συμβιβασμού, λοιπόν για τι αιτιολογικές σκέψει και για αυτού του συμβιβασμού θέλουμε να υποστηρίξουμε ότι για τις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας δεν πρέπει να θεωρούνται ως περιορισμοί. Ακόμη και αν φυσικά θέλουμε να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την δράση τους. Στο συμβιβασμό Β τώρα τι έχουμε. Από ό,τι κατανόησα θα υπάρξει μία τροποποίηση ή βελτίωση γλωσσικού χαρακτήρα. Τώρα τι λέμε. Λέμε και οι πέντε οδηγίες θα πρέπει να ε, επανεξεταστούν για να παράσχουμε κτλ. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα επανεξεταστούν και θα αναθεωρηθούν. Και η κυρία Χάκιν από ό,τι κατάλαβα θα υπο... καταθέσει μια προφορική τροποποίηση για την καλύτερη διατύπωση. Αλλά το περιεχόμενο δεν θα αλλάξει, η ουσία δεν θα αλλάξει. Και είμαι σχεδόν βέβαια ότι μπορούμε να δεχθούμε αυτές τις ε, γλωσσικές ή διατυπωτικές βελτιώσεις. Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί είναι τεχνικού χαρακτήρα περισσότερο. Μπορούν να γίνουν δεκτές σε μεγάλο βαθμό, γίνονται δεκτές από τους τεχνικούς επαΐοντες, ε, τους πραγματογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι λοιπόν από ό,τι γνωρίζω δεν θα υπήρχαν κάποια προβλήματα, δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα με αυτές τις προτάσεις. Αυτά για αύριο που ελπίζω ότι πραγματικά μπορούμε να καταλήξουμε στη συμφωνία πρώτης ανάγνωσης και να ολοκληρώσουμε. Και ελπίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το αίτημα. Από πλευράς μου θέλω μόνο να ευχαριστήσω λοιπόν τους σκιώδεις εισηγητές ε, που ήταν πολύ δραστήριοι και συνεργάστηκαν πολύ για αυτό το θέμα μαζί μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σάρι. Πολύ καλά φαίνονται ότι πάνε τα πράγματα. Να δούμε αν θα παραμείνουν τόσο καλά. Όλοι οι Κρίστενσεν, ε, σκιώδης εισηγητής από πλευράς ε, σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ επίσης και την εισηγήτρια για την πολύ καλή καλή συνεργασία που είχαμε. Χαίρομαι πρέπει να πω για το ότι υπήρξε ανταπόκριση στα αιτήματά μας και οι δικές μας σκέψεις και προτάσεις κατέληξαν στους συμβιβασμούς. Πρώτον, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ασφάλεια και η προστασία της υγείας ε, στον χώρο εργασίας δεν πρέπει να θεωρείται επιβάρυνση και δαπανηρή διαδικασία και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για πρόσχημα, προσχηματικά ώστε να μην προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο διασφαλίζουμε και πρέπει να διασφαλίζουμε ώστε θεμελιώδε δικαίωμα. Τονίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες ειδικέ, ιδιαίτερε ομάδε που εκτίθενται σε ειδικού κινδύνους. π.χ. χημικέ ουσίε. Αυτό αφορά επίσης και κομμωτές για παράδειγμα και κουρίς που έχουν να κάνουν με επικίνδυνες ουσίες και που πολλές φορές εργάζονται χωρίς να έχουν πληροφορηθεί ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούν στο επάγγελμά τους. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια για το ότι προσπάθησε να ανταποκριθεί σε αυτά τα θέματα στις, ε, στα αιτήματά μας ώστε να καλύπτονται οι εργαζόμενοι όπως πρέπει σωστά. Πρόεδρος, ευχαριστώ αγαπητέ Όλε για την flexicurity εσείς ε, για την φιλελεύθερη ομάδα η κυρία Χάρκιν, αλλά από πλευράς Φιλ Μπέγκε θα λάβει τον λόγο ο ίδιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ Χαίρομαι για το ότι είναι δυνατόν. Ομιλώ τώρα να εξ ονόματος της συναδέλφου. Θέλω να ευχαριστήσει το, την εισηγήτρια για την εξειδικευμένη σε βάθο και αποτελεσματική δουλειά για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Παρότι είναι ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα, η επικοινωνία τη κυρία Χάρκιν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαγνώσει αυτή την υποστήριξη που υπάρχει για αυτή την τάση όπω παρουσιάστηκε. Για την ορολογία σε σχέση με την κυρία Χάρκιν όπω πιστεύει ότι πρέπει να δικαιολογείται και να συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο για το δεύτερο τμήμα θα ήθελα να ζητήσει από την εισηγήτρια η κυρία Χάρκιν για τις πέντε αυτές οδηγίες που θα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδική εξέταση αναθεώρηση. Αν θα είναι διαρκώς υπό εξέταση τότε θα έχουμε μια διαρκή ε, υποεξέλιξη διαδικασία και θα δημιουργείται ανασφάλεια ή αβεβαιότητα. Τι συμβαίνει με το ένα ή άλλο έγγραφο και ποια μορφή θα έχει το τελευταίο έγγραφο αν υπάρχει διαρκώς μια αναθεώρηση σε εξέλιξη. Η Άντε θα προτιμούσε μια πιο διαθρωμένη η δομημένη προσέγγιση, δηλαδή να υπάγονται σε περιοδική αναθεώρηση και επανεξέταση και όχι σε διαρκή αναθεώρηση και επανεξέταση. Και σε σχέση με τις τροπολογίες προσβλέπει η κυρία Χάρκιν στο να διεξαχθεί η ψηφοφορία αύριο επ' αυτών. Ευχαριστώ. Άλλοι ευρωβουλευτέ θέλουν να παρέμβουν. Η Σάρη στο τέλος θα παρέμβει. Δεν υπάρχουν άλλοι. Η Επιτροπή. Θα ήθελε η Επιτροπή να τοποθετηθεί παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις τροπολογίες σας. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουν να υπογραμμίσουν ότι οι τροπολογίες σας έχουν να κάνουν κυρίως με τη γράμμιση στην ορολογία άλλες διευκρινίσουν κάπως Θέλετε επίσης να προσθέσουμε κάποιες ε, άλλες ε, κατηγορίες και τις οδηγίες να είναι τέτοιες που να προσαρμόζονται στην πρόοδο. Θέλω όμως εδώ να σας πω ότι οι τροπολογίες 10 και 11 μας απασχολούν κάπως γιατί εμείς θεωρούμε ότι δεν φτάνει να αναφερόμαστε στις υποκατηγορίες 1α ή 1β πρέπει να αναφερόμαστε και στην κατηγορία 1, γιατί η κατηγορία 1 καλύπτει επίσης περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δυνατότητα υπό κατηγορίας 1α ή 1β, για ορισμένες περιπτώσεις ουσιών δηλαδή. Συνεπώς πιστεύουμε ότι εδώ θα έπρεπε πρώτον να μην λέμε 1α και 1β, αλλά να λέμε 1α ή 1β και επιπλέον για τις τροπολογίες 23 και 24 κάποια τμήματα των τροπολογιών αυτών ίσως να μην έχουν άμεση σχέση με το πλαίσιο της παρούσας πρότασης που είναι οι πέντε οδηγίες. Ωραία. Ευχαριστώ για την Επιτροπή και στο τέλος η κυρία Συγήτρια να ολοκληρώσει. παρακαλώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τα σχόλιά της και είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια του τριμερή διαλόγου. Συμφωνώ απόλυτα ότι η διατύπωση περιοδική αναθεώρηση είναι προτιμότερη, οπότε θέλω να ζητήσω από τη Γραμματεία θα υπάρξει τέτοια τροπολογία αύριο Εντάξει, θα μπορέσουμε δηλαδή να συμφωνήσουμε όλοι, ε, γιατί νομίζω και εγώ ότι στα αγγλικά η διατύπωση έτσι είναι προτιμότερη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Νικτερινή εργασία προβλέπετε ότι θα γίνει, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Αύριο θα ψηφίσουμε γι' αυτό, Σάρι. Καλό είναι λοιπόν σήμερα να δοθεί αυτό στη γραμματεία ώστε να προετοιμαστεί. Το επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη που έχουμε είναι το σημείο 5 λοιπόν εφαρμογή της οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Εισηγητής ο φίλος μας Άνταμ Κώσα. Άνταμ έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα αναφερθώ στις συμβαστικές τροπολογίες. Υπάρχουν επτά συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε υποβάλει. Την προηγούμενη φορά είχαμε μια εξαιρετική συνεδρίαση με τους σκιώδεις εισηγητές. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ θετικό, μπορέσαμε πολύ ανοιχτά να συζητήσουμε τις απόψεις μας και εντοπίσαμε ποιες είναι οι τροπολογίες αυτές οι οποίες μπορεί να γίνουν συμβιβαστικές. Νομίζω ότι οι περισσότερες από τις πολιτικές ομάδες είναι ικανοποιημένε με τις συμβαστικές αυτές προτάσεις. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολο να καταλήξουμε σε μία λύση με την οποία να συμφωνούν όλοι. Υπάρχει πάντως μία προβληματική συμβαστική τροπολογία. Στην δικιά μου αρχική τροπολογία είχα προσπαθήσει να διατηρήσω την ισορροπία. Οι πολιτικές ομόδες ελπίζω τελικά να το δεχτούν. Γιατί πώς κάνεις διαφοροποίηση και που μιλάμε για τις διακρίσεις, έτσι. Φαντάζομαι ότι είναι η τροπολογία D. Πρόκειται για την διάκριση σε βάρος. Στους χώρους εργασίας κλπ. Μια στιγμή να βρω τα χαρτιά μου, Λέω μιλητής. Στις συμβαστικές τροπολογίες προσπάθησα να καταδείξω ότι δεν μιλάμε μόνο για την τροπολογία 70 του 2000 συνολικά οι συμβαστικές τροπολογίες όλες και κάθε μία χωριστά βασίζονται μόνο και αποκλειστικά στην οδηγία 78-2000 αλλά για την οδηγία αυτή ελπίζουμε να μπορέσουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέξουν, τι μελέτες πρέπει να εκπονήσουν. Το ίδιο ισχύει και για την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά είχα να πω και τώρα περιμένω τις δικές σας παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστώ θερμά, Άντα. Για τους σκιώτες συζητητές, Κυβέτη η πρώτη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κώσα θερμά για την επικοδομητική συνεργασία από πλευράς του. Είχαμε μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό κλίμα εργασίας κατά τις επαφές και συζητήσεις μας. Από τη δική μας πολιτική ομάδα θα θέλαμε για τον συμβιβασμό Α να παρατηρήσουμε το εξής. Το τελευταίο τμήμα αυτής της τροπολογίας, τροπολογίας 37 δηλαδή, δεν θα έπρεπε να ενταχθεί στο συμβιβασμό. Γιατί αυτή η τροπολογία αποσύρθηκε ουσιαστικά. Ή εμεί θα την αποσύρουμε, εν πάση περιπτώσει. Ο συμβιβασμός Α λοιπόν παραμένει ως έχει και ως προβλέπεται αυτή τη στιγμή μόνο αυτή η τροπολογία 37 που συμπεριλαμβάνεται πρέπει να διαγραφεί να αποσύ... γιατί εμείς θα την αποσύρουμε. Μετά περνάμε στον συμβιβασμό ε, τον πέμπτο. Δεν μπορούμε να τον υποστηρίξουμε ως έχει στη διατύπωσή του τώρα αυτό το συμβιβασμό. Ως έχει στη διατύπωσή του δεν μπορούμε να τον δεχτούμε και να τον υποστηρίξουμε. Τι αναφέρεται ουσιαστικά σε αυτή την πρόταση τροπολογίας. Λέγεται ότι απουσιάζουν στοιχεία. Δεν είναι ίσως διαθέσιμα τα στοιχεία τα οποία απουσιάζουν λόγω προβλημάτων κτλ. Που όμως είναι σημαντική υπόθεση. Λένε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Εμείς θεωρούμε κάτι διαφορετικό, πιστεύουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλά στατιστικά στοιχεία για αυτό το θέμα, δεν απουσιάζουν. Πέρα από αυτό υπάρχουν ευρωπαϊκά όργανα και ευρωπαϊκά, ο ευρωπαϊκοί οργανισμοί που έχουν συντάξει πολλά τέτοια στοιχεία που έχουν συλλέξει και έχουν συντάξει και εκθέσεις για αυτό το θέμα και έχουν διατυπώσει και απόψεις, γνωμοδοτήσεις με στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι αξιόπιστα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο λέγεται ότι απουσιάζουν αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το τμήμα εκείνο αυτού του συμβιβασμού που αφορά την τροπολογία 33 και απευθύνομαι άμεσα τώρα προς τον εισηγητή, Λοιπόν, ήδη σας το γνωστοποίησα ποια είναι η άποψή μας γι' αυτό, αλλά θα ήθελα δημόσια να το επαναλάβω και να το τονίσω. Τροπολογία 33 λοιπόν. Εμείς θα είμαστε υπέρ ώστε ξεχωριστά να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Ναι, μεν εντάχθηκε στο συμβιβασμό όμως, μια και εμείς πιστεύουμε ότι η πλειοψηφία αυτή αυτής της συμβαστικής τροπολογίας δεν μπορεί να γίνει δεκτή από εμάς, επιφυλασσόμεθα την 33 να ζητήσουμε να ψηφιστεί χωριστά. Και πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες που δεν καλύπτονται από τους συμβιβασμούς, από τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Τι κάνουμε λοιπόν. Υποστηρίζουμε μεν αυτές τις τροπολογίες, αλλά θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική έκθεση και ελπίζουμε ότι στην ψηφοφορία δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Ευχαριστούμε συνάδελφε για την άλλη τώρα. Σύρι παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μου καταρχήν στηρίζει την οδηγία αυτή. Φυσικά πρέπει να επικαιροποιηθεί, να εξυγχρονιστεί. Και γι' αυτό ευχαριστούμε τον κύριο Κώσα που συνεργάστηκε πολύ καλά με τους κοιόδες συζητητές και αυτά που μας παρουσιάζονται είναι 55 τροπολογίες. Φτιάξαμε 7 συμβαστικές τροπολογίες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να στηρίξουμε, αλλά υπάρχουν και τροπολογίες που δεν είναι συμβατές με τη δική μας θεώρηση. Δυστυχώς. Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε σε δύο κατηγορίες τροπολογίες είναι κάποιοι οι οποίοι εξακολουθούν να θέλουν να εξηγήσουν την απόψή τους ή να ενταχθούν στην οδηγία πέντε τομείς. Πέντε βιβλίων τομείς. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όμως δεν είναι αποδεκτά. η άλλη κατηγορία, αντί για αναδιατύπωση, μιλάει για επικαιροποίηση απόλυτα δικαιολογημένη. Η πλειοψηφία αυτών των τροπολογιών μπορούμε να, μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμά την πλειοψηφία της δεύτερης κατηγορίας τροπολογιών. Ε, στηρίζουμε το 85% των τροπολογιών. Η τροπολογία F. Δεν την καταλαβαίνουμε. Επιθεώρηση στους χώρους εργασίας. Νομίζουμε ότι είναι περιττό αυτό. Δεν στηρίζουμε αυτόν τον συμβάσμα, τον συμβάσμο F. Λοιπόν, εν συνεχεία. Μπορούμε να στηρίξουμε την αιτιολογική, αιτιολογική σκέψη παριθμών 1. Το πρώτο τμήμα αυτή της αιτιολογική σκέψης είναι απόλυτα αποδεκτό. Αλλά το δεύτερο τμήμα, υπό τη μορφή προφορική τροπολογία. δεν είναι αποδεκτό. Κατά κανόνα, η δουλειά του κυρίου Κώσα μαζί με τους σκιώδες εισηγητές ε, ήταν πολύ καλή, με κάποιες εξαιρέσεις. Επομένως μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση. Σα ευχαριστώ θερμά. Για τους πράσινους η Ελίζα Μπεξουρέντα παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση ουσιαστικά. Και αυτό γιατί. Διότι η ιδέα ήταν σε αυτή την έκθεση την έκθεση ιδέα πρωτοβουλία να τη συντάξουμε προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέσει και υποβάλει τη δική τη έκθεση που σύμφωνα με τον κανονισμό σύμφωνα με την οδηγία είναι υποχρεωμένη να συντάξει. Αυτή είναι η ιδέα δηλαδή, να δώσουμε ερεθίσματα εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για την επίσημη έκθεση που θα αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να συμπεριληφθεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απογοητευτική αυτή η έκθεση. Μας απογοητεύει επειδή δεν αξιολογεί όλους τους λόγους ισότιμα. Πώς δηλαδή στην οδηγία διαδραματίζουν ένα ρόλο και ποια επίπτωση έχουν. Και ουσιαστικό ήταν στις δικές μας τροπολογίες να αποκαταστήσουμε την ισορροπία που αρχικά δεν ήταν δεδομένη, δεν υπήρχε. Στόχος είναι φυσικά εδώ και πάλι το σύνολο της πολιτικής κατά των διακρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε λίθαργο να την αναζωογονήσουμε και να δώσουμε κίνητρα σε αυτή την πολιτική κατά των διακρίσεων. Αυτοί ήταν οι λόγοι με τους οποίους ξεκινήσαμε. Δεν τα καταφέραμε όμως να εκπονήσουμε αυτά τα κίνητρα και αυτά, <clears throat> αυτές τις θετικές ιδέες. Υπήρξαν κάποια κολλήματα, κάποιες ε, κάποια προβλήματα. Επί μεγάλο χρόνο, επί μεγάλο χρονικό διάστημα εργαστήκαμε για τις συμβαστικές τροπολογίες και μπορούμε να πούμε όπου εκεί όπου δεν έχουν όλες ισότιμα εξεταστεί έχουμε πρόβλημα εκεί όπου δεν αξιολογούνται όλα τα θέματα ισότιμα κυρίως έχουμε ένα πρόβλημα ότι σημαντικά θέματα όπως η gender identity η ταυτότητα φύλου που σε σχέση με την απόφαση των συντονιστών έπρεπε να ενταχθεί στην έκθεση σε ξεχωριστό σημείο δεν έγινε αυτό. Και δεν έγινε αυτό το οποίο από πλευρά συντονιστών είχε προβλεφθεί. Πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση ίσως για να το ρυθμίσουμε το θέμα. Ίσως με επιστολή της Προέδρου Πάντως στην έκθεση δεν συμπεριλήφθηκε τίποτα από αυτά που είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν και υπάρχει αυθεντικό κενό λοιπόν, υπάρχει αυθεντικό χάσμα σε σχέση με την εντολή που είχαμε δώσει. Για την, ε, τον συμβιβασμό, την λύση για το, την πρόταση α με την ε, απόσυρση της προσθήκης, αν συμβαίνει αυτό μπορούμε να δεχτούμε και να υπεψηφίσουμε αυτόν τον συμβιβασμό γιατί δεν θα δεχόμαστε τη συμπλήρωση αυτών, την προσθήκη αυτών. Για, ήθελα να δώσω το, ε, το δίκιο ε, στα όσα αναφέρθηκαν από πλευρά συναδέλφου ότι αναφέρθηκε λέει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν διακρίσεις. Έχουμε όμως τέτοια στοιχεία και μια τέτοια μελέτη από, την, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και είναι λάθος να υποστηρίζει κανείς ότι δεν υπάρχουν λέει τέτοιες διακρίσεις και στοιχεία για τέτοιες διακρίσεις με βάση την σεξουαλική ταυτότητα. Δεν αληθεύει αυτό καθόλου μάλιστα. Και γι' αυτό μπορούμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κανένα τρόπο. Άλλους συμβιβασμούς τους δεχόμαστε. Και σε σχέση με την εισηγήτρια της το έχουμε ήδη γνωστοποιήσει αυτό. Για μας εξαρτάται λοιπόν η υπόθεση από το ποιες τροπολογίες θα περάσουν σε σχέση με αυτή την έκθεση. Για να δούμε αν στο τέλος θα υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση ή όχι. Δεν είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με το πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Αν με καλές τροπολογίες, ιδιαίτερα με τις τροπολογίες από πλευρά συναδέλφου Τιβέτη αποδυναμωθεί η έκθεση, τότε θα επιφυλαχθούμε αν θα υπερψηφίσουμε ή όχι. Θα το δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ελίζαμπετ για τα σχόλιά σου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποιο από την Επιτροπή. εσεί παρακαλώ. Εσείς παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Πέτρα Σότα από την Επιτροπή. Προέρχομαι από το τμήμα που είναι υπεύθυνη, την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Μπορώ και πάλι να σας ξαναπώ αυτό το οποίο από πλευρά συναδέλφου αναφέρθηκε, ότι δηλαδή αυτή η έκθεση μέχρι τα τέλη του έτου θα υποβληθεί, θα κατατεθεί θα δημοσιοποιηθεί και θα αναφέρεται και στις δύο οδηγίες, τη 2043 για τη, τη διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την φυλή ή την εθνότητα και την 2078 που ε, έτσι θα καλύπτει και τις δύο αυτές, ε, τα δύο αυτά σκέλη και θέτουμε το κέντρο βάρους ε, στις διακρίσεις λόγω ηλικίας. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά κυρία Σότα. Και τώρα θα λάβει τον λόγο Άνταμ κόσα να συνοψίσει για μια όχι τόσο απλή από ό,τι βλέπουμε έκθεση. Κύριε Κόσα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις τους που με καθησύχασαν. Προσπάθησα να λάβω υπόψη τη γνώμη όλων των πολιτικών ομάδων όσο μπορούσα. Φυσικά δεν μπορούσα να το κάνω αυτό 100% και δεν μπορούσα να ικανοποιήσω όλους 100% αλλά νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες υποστηρίζουν το συμβαστικό πακέτο. Για την ε, συμβαστική τροπολογία A ε, δεν έχω πρόβλημα να συμφωνήσω με τους σοσιαλιστές αλλά Η έκφραση ακραίων πεπιθήσεων είναι βασικό θέμα. Γι' αυτό βρήκα τη λύση που βρήκα στην τροπολογία α, α, ε. Για τροπολογία ε, ε. Το κοίταξα με τους συναδέλφους. Η οδηγία 78 καθώς 2000 καλύπτει διάφορες ομάδες, όχι όμως Δεν υπάρχουν όμως μελέτες ή στατιστικά στοιχεία για όλες τις ομάδες στη διάθεση της Κομισιόν. Δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία, Φερρυπίν, για τις διακρίσεις που υφίσταται κανείς λόγω θρησκείας. Συμφωνώ λοιπόν με τους συναδέλφους που είπαν ότι θα πρέπει να αναφέρουμε τις μελέτες και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ναι, όντως θα πρέπει να αναφερθούν. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε, να τονίσουμε πού υπάρχουν ανελειπή στοιχεία ή όπου δεν υπάρχουν, που δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, στατιστικά και μελέτες. Έχουμε ένα πακέτο συμβαστικών τροπολογιών και πιστεύω ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων θα υποστήριξε αυτό το συμβαστικό πακέτο. Σε ό,τι αφορά τις χωριστές ψηφοφορίες. Για να δούμε τι θέλετε ακριβώς. Μιλούσατε για την τροπολογία 37. Οι σοσιαλιστές δεν θέλουν να... Ε, η τροπολογία 37 να συμπεριληφθεί και θέλουν να ε, χωριστή ψηφοφορία ή μάλλον ψηφοφορία κατά τμήματα ε, για την 37 και αν 37 δεν ρυθμιστεί, τότε δεν θα ψηφίσουν τροπολογία, τη συμβαστική τροπολογία Α. Αυτό για να το καταλάβω καλά. Ε, κατά τα άλλα σας ευχαριστήσω όλους για την επικοδομητική σας συνεργασία. Ίσως Μου είπαν δεν υπάρχει διερμηνία λέει. Τι συμβαίνει. Δεν ήταν σαφές για την τροπολογία 37 που ήταν ε, σε σχέση με την ψήφιση θα αποσυρθεί από το συμβιβασμό η 37. Εντάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Εντάξει, ένα πρόβλημα λιγότερο, Άνταμ. Εντάξει, λοιπόν, καλό θα ήταν να τεθείτε σε επαφή οι δυο σας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε χωρίς προβλήματα αύριο. Ευχαριστώ θερμά. Πολύ καλά. Περνάμε λοιπόν στη συνέχεια. Ε, αναγκαστήκαμε να τροποποιήσουμε την ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο 8 τώρα της ημερήσιας διάταξης. Birgit Zippel έχει τον λόγο. Το θέμα είναι ΚΑΣ 2020 για μια ισχυρή ανταγωνιστική βιομηχανία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία. Έχει τον λόγο, Μπίρκιν, να δούμε για τι τροπολογίε τι γίνεται. Ευχαριστώ. Έγκαιρα λοιπόν ήρθα στην αίθουσα για να δούμε αυτό το θέμα. Πολύ καλά. Πρόκειται εδώ λοιπόν για μια γνωμοδότηση τη δική μα κοινοβουλευτική επιτροπή για το έγγραφο ΚΑΣ 2020 αυτοκίνητα 2020. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές Είχαμε μια συνεδρίαση όπου στα ουσιοθέστερα θέματα, νομίζω 7 συμβιβαστικές τροπολογίες ήταν αυτές, συμφωνήσαμε επ' αυτών. Υπάρχει συνένεση ιδιαίτερα για το ότι όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, είναι σημαντική αυτή. Τα αυτοκίνητα είναι πολύ σημαντικά για την κινητικότητα των ανθρώπων στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα της αυτοκίνησης με, μεγάλη έρευνα και μεγάλη ανάπτυξη σημειώνεται και δεδομένων των διαρκών προκλήσεων με μεγάλα, μικρά αυτοκίνητα, διασφάλιση και διαφύλαξη των πόρων και το θέμα της ανταγωνιστικότητας εδώ καλύπτεται και το θέμα των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων σε αυτή τη βιομηχανία. Πολύ σημαντικά σημεία που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη ως Επιτροπή Απασχόλησης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για μας. Ίσως τώρα από πλευρά μου να, δούμε τις, να δω τις τροπολογίες σύντομα και να σας επεξηγήσω. Στο συμβιβασμό Α υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά τη σπουδαιότητα του τομέα της αυτοκίνησης συνολικά. Και αναφέρουμε και αυτό κιόλας που στο συμβιβασμό Β για άλλη μία φορά λέμε και εξηγούμε ότι σε, αυτή την, σε αυτό τον τομέα γίνεται πολύ μεγάλη καινοτομία. Σημειώνεται μεγάλη καινοτομία και είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε, να γίνουν οι επενδύσεις και είναι αυτό σημαντικό και για την απασχόληση στην Ευρώπη να βρισκόμαστε ως πρωτοπόροι, να είμαστε οι πρώτοι που θα εισαγάγουμε την καινοτομία για να διασφαλίσουμε τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι άλλο. Έχουμε επίση ένα συμβιβασμό, μια συμβαστική τροπολογία όπου πρόκειται για τις διαρθρωτικές προσαρμογές Και πάλι και πάλι για το ζήτημα πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε στο να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις με τον καλύτερο τρόπο και να μεριμνήσουμε ότι οι αναγκαίες προσαρμογές <clears throat> δεν θα οδηγήσουν στο να υπάρχουν αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη ή με άλλα λόγια αυτές οι επιπτώσεις να τηρηθούν, να κρατηθούν σε ένα ελάχιστο επίπεδο και επισημαίνουμε εδώ και το θέμα <clears throat> της κατάρτισης και εκπαίδευσης και των σχεδίων και προγραμμάτων για τους εργαζόμενους ώστε να είναι οι εργαζόμενοι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες ε, προκλήσεις. Διαθροτικές μεταβολές και αλλαγές. Φυσικά στο συμβιβασμό Δέλτα, στον, στο στον τέταρτο συμβιβασμό γίνεται λόγος για τον ρόλο του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη, κλείσιμο βιομηχανίας ή σημαντική μείωση των εργαζομένων σε κάποια βιομηχανία, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης να μπορεί έγκαιρα νωρίς να δρά και να υποστηρίζει με ειδικά μέτρα τους απασχολούμενους σε αυτές τις βιομηχανίες. Και σε όλα τα κράτη-μέλη αυτή η δυνατότητα να προβλέπεται ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε βάθος από αυτά αν είναι ανάγκη. Δεδομένων όλων αυτών των προκλήσεων υποστηρίζουμε επίσης την ίδρυση ενός Skill Council θέλουμε όλοι να συνέρχονται σε μια πλατφόρμα για να δουν, να βλέπουν ποιες προκλήσεις υπάρχουν για την εκπαίδευση, κατάρτιση, πώς μπορούν να διοργανωθούν οι αναγκαίες εκείνες ε, εκδηλώσεις για την κατάρτιση και επιμόρφωση και εκπαίδευση των ε, εργαζομένων, να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε μια τέτοια πλατφόρμα, να δούμε τι μπορούμε να διοργανώσουμε. Αναφέραμε ήδη το Ταμείο παγκοσμιοποίηση, για το Κοινωνικό Ταμείο ως μακροπρόθεσμο μου χαρακτήρα μέτρο, είναι σημαντικό στον τομέα της εκπαίδευσης ε, να παρεμβαίνουμε ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ε, νέων τεχνολογιών όσον αφορά τους απασχολούμενους, τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό και να είμαστε στο ύψος των, περιστάσεων στην ε, ε, τροπολογία G λέμε πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε ως συμπληρωματικό μέσο στην αγορά εργασίας αυτή τη δυνατότητα στις εθνικές ε, οργανώσεις και όργανα να συμβουλεύουμε τους εργαζόμενους πώς μπορούν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους να τις αναπτύξουν περαιτέρω, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης πλήρους χρόνου, δηλαδή πλήρους απασχόλησης και να μπορούν έτσι να χρηματοδοτηθούν αυτές οι, προ... οι εκδηλώσεις και να ε, μπορούν οι εργαζόμενοι να τις ε, χρησιμοποιήσουν, οι ε, ε, εργοδότες να τις χρησιμοποιήσουν αυτές τις εκδηλώσεις για να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Για την τροπολογία Α είμαστε η Επιτροπή Απασχόλησης και το θέμα του labeling των συσκευασιών και ετικετών υπάρχει ένα συμπλήρωμα ότι καλό θα ήταν να υπάρχει μια ετικέτα για το διοξίδιο του άνθρακα. Σε κάποια κράτη-μέλη το έχουμε αυτό. Ήταν όμως επίμαχο αν ανήκει σε αυτό το πλαίσιο ή όχι αυτή η πρόταση. προταση εμείς θα θέλαμε να προτείνουμε τον συμβιβασμό Α να τον θέσουμε σε ψήφιση, σε ψηφοφορία ως έχει. Το σημείο για το διοξίδιο του άνθρακα να είναι προσθήκη σε αυτό τον συμβιβασμό Α. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε τώρα στις εκθέσεις των σχεδόν εισηγητών. Για το ΕΛΚ ήταν η Βερονίκα. Λόπες, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια, την κυρία Σίπελ. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ότι συνεργαστήκαμε καλά μαζί και ότι καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτές τις συμβατιστικές προτάσεις που θα στηρίξει το ΕΛΚ. Αφαιρέθηκαν κάποια σημεία τα οποία ήταν περίπλοκα για όλους και έτσι πιστεύω ότι καταλήξαμε σε ένα κείμενο το οποίο μας ικανοποιεί όλους. Την αυτοκινητοβιομηχανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορες περιφέρειες και τη δικιά μου, όπου είναι κάτι αναγκαίο για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Πρέπει επίσης εμείς η Επιτροπή Απασχόλησης να υπογραμμίσουμε τα θέματα της ασφάλειας και της ποιότητας. Είναι επίσης θετικό να στοιχηματίσουμε για, στον τομέα αυτό προκειμένου να γίνει πιο πράσινος και να προστατεύει καλύτερα το περιβάλλον στο μέλλον. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε η γιατί συμφωνώ μαζί της με όλες τις συμβαστικές της προτάσεις που συζητήθηκαν στην ομάδα και μας βρίσκουν σύμφωνους. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου, για παράδειγμα, προκειμένου οι εργαζόμενοι να καταρτίζονται κατάλληλα και έτσι να προλαμβάνουμε τις ανάγκες που θα έχει ο τομέας στο μέλλον. Έπειτα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση να στηρίζουμε τους εργαζόμενους εκείνους οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω αναδιάρθρωσης. Και όταν μιλάμε για αναδιάρθρωση, η συμβαστική τροπολογία ΓΑΜΑ πολύ σωστά αναφέρεται σε στρατηγικές υπέρ του πληθυσμού προκειμένου να προκαταλαμβάνουμε τις μελλοντικές ανάγκες του τομέα και να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα αναδιάρθρωσης. Είναι κάτι το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και στην έκθεση ΣΕΡΚΑ. Η γνωμοδότηση αυτή λοιπόν μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή και ελπίζω ότι θα την εγκρίνουμε χωρίς καμιά δυσκολία. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, θερμά. Μπάνιαν για τους ε, φιλελεύθερους, παρακαλώ. Φιλ Μπάνιαν. Ευχαριστώ, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για ό,τι έκανε. Συμφωνούμε. Είναι μια πολύ θετική γνωμοδότηση αυτή. Η υπόθεση, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εκλογική μου περιφέρεια ιδιαίτερα, διότι έχουμε τεράστια δυνατότητα απασχόλησης και 1.700 νέες θέσεις μπορούμε να έχουμε από μια ε, πρωτοβουλία design. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε και ένα εργοστάσιο που θα φτιάχνει μηχανές 10.000 θέσεις απασχόλησης είχαμε τα τελευταία χρόνια στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια και μόνο. Και γνωρίζω επίσης πάρα πολύ καλά ότι χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια στην περιφέρειά μου για έρευνα. για να βελτιωθεί και η ασφάλεια και η εξοικονόμηση καυσίμων και η εξοπιστία γενικά των προϊόντων τους. Συνεπώς στηρίζουμε όλες τις τροπολογίες. Δεν λέω τα πάντα σε όλες, πάντως τις συμβαστικές ναι. Οι συμβαστικές έχουν λάβει υπόψη τις δικές μας τις ανησυχίες και οι άλλες ομάδες κάνανε επικοδομητικές προτάσεις. Η συμβαστική Α είναι ιδιαίτερα θετική και τονίζει αυτά που είπα και εγώ νωρίτερα για τις δυνατότητες που έχει η αυτοκινητοβιομηχανία και η εφηπίσεις που αναφέρεται στην κατάρτιση και επανακατάρτιση των εργαζόμενων. Πρέπει να φροντίσουμε για ευκαιρίες στον τομέα αυτό. Στις συναντήσεις με τους κοιόδες και με τις δικές μου προσπάθειες καταφέραμε να κρατήσουμε θετική τη γνωμοδότηση αυτή, γιατί υπήρχε κάποια άποψη που έλεγε ότι έπρεπε να φαίνεται ότι είναι σε ύφεση η βιομηχανία και τέτοια. Εγώ δεν συμφωνούσα, δεν ήθελα να υπάρξει μια τέτοια απόχρωση στη γνωμοδότηση, έπρεπε να βλέπουμε τη θετική πτυχή, μια που μιλάμε για ανάκαμψη, για τις δυνατότητες που έχει η αυτοκινητοβιομηχανία. Υπάρχει μια επιτυχία και αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία να είναι ανταγωνιστική παγκοσμίω και να αποτελέσει μια ευρωπαϊκή success story. Ευχαριστώ πολύ Φίλιπ. Δεν θέλει κάποιο άλλο να παρέμβει, έτσι. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τον λόγο. Έχω την κυρία Κουνόβα, σωστό αυτό. Εσεί είσαστε εδώ παρούσα. Κουξόβα. Uh, Από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων σας ευχαριστούμε για τα πολύ επικοδομητικά σας σχόλια. Δεν έχουμε ιδιαίτερα άλλα σχόλια να προσθέσουμε όμω. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κούξοβα. Σωστό το όνομα. Μπίργκιτ, για να ολοκληρώσει έχεις τον λόγο. Και αύριο θα ψηφίσουμε Μπίργκιτ, εντάξει. Πες μας τα σχετικά. Αύριο θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για άλλη μια φορά για αυτή τη συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Μπένιον που ανέφερε τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης για άλλη μια φορά. Διότι πραγματικά δεν θέλουμε κάποια αυτοβιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία να έχουμε στην Ευρώπη, αλλά θέλουμε να είμαστε πρότυπο και υπόδειγμα για όλους τους άλλους και για τους κινητήρες και για την κατανάλωση καυσίμου και τα λοιπά, να είμαστε πρωτοπόροι και για το θέμα των υλικών που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Γι' αυτό συνολικά με τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και τις τροπολογίες βρισκόμαστε σε σωστή πορεία. Ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε καλή συνεισφορά και καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αύριο η ψήφιση, η Ήτρε θα ακολουθήσει στις 17 Οκτωβρίου από πλευρά Ήτρε. Ελπίζουμε ότι πολλά θα εντάξει η Ήτρε από αυτά που αύριο θα εγκρίνουμε εμείς. Αυτό είναι το σημείο 8. Περνάμε στο 9. Η συγγήτρια είναι παρούσα, η κυρία Φρανσουάζ Καστέξ, για το θέμα σε σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φρανσουάζ, έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε είχαμε ειδωθεί την τελευταία, την περασμένη εβδομάδα, όταν ανταλλάξαμε απόψεις. Υπήρχαν ε, σε πολλά σημεία σύγκλησης, Υπήρχαν σε πολλά σημεία σύγκληση μεταξύ των Ευρωβουλευτών ε, στο κείμενο που σας υπέβαλα. Αυτές, ε, αυτά τα σημεία σύγκληση επιβεβαιώθηκαν με την εκπόνηση των συμβαστικών τροπολογιών. Έχουμε 8 συμβαστικές τροπολογίες Ουσιαστικά δηλαδή το σύνολο της νομοδότησης καλύπτεται από αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Μας επέτρεψαν να βρούμε σημεία σύγκληση σε όλες οι πολιτικές ομάδες. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αφορούν Τι επιφυλάξει κυρίως που έχουμε από πλευρά μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού όλος ιδιαίτερος, ότι το δίκαιο ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει τις επενδύσεις στους στρατηγικούς τομείς. Θα πρέπει να διατηρήσει τις κοινωνικές πολιτικές και να λαμβάνει υπόψη τις, ε, τα όσα επιτάσσει στο άρθρο 9 και στο άρθρο 14, καθώς και στο πρωτόκολλο 26 για τις ε, υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, συνθήκη της Λισαβόνας. Οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος να μην ε, εντάσσονται στον ε, έλεγχο ανταγωνισμού, γιατί δεν στραβλώνουν τον ανταγωνισμό, αλλά πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται σε μία συγκεκριμένη ε, εθνική επικράτεια και επομένως δεν υπάρχει εδώ πέρα θέμα διασυνοριακού ανταγωνισμού. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν να προσθέσουν κάτι, αλλά μπορούμε νομίζω να, να ψηφίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση αύριο χωρίς κανένα πρόβλημα και πιστεύω ότι θα υπάρξει ευρία πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Φρανσουάς. Ευχαριστώ. Α, Κάζα, παρακαλώ για τον λόγο. Από πλευρά του Έλκ, Σκιώδη. παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω υπόθηκε, δεν υπήρξαν προβλήματα, δεν ήταν επίμαχη αυτή η έκθεση. Ξέρετε ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι σημαντική για την ε, εσωτερική αγορά. Είναι σημαντική για να ισχυθεί και να γίνει πιο βιώσιμη η εσωτερική αγορά. Φυσικά η, πολιτική ανταγωνισμού βοηθάει τους καταναλωτές στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να τους βοηθάει μάλλον και να προστατεύονται καλύτερα οι καταναλωτές. Είμαι ικανοποιημένος από τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε. Κυρίως συμφωνώ με την έμφαση που δίδεται στην προστασία των καταναλωτών. Εκεί που ζητάμε τη μείωση της απάτης στα φορολογικά ζητήματα, με βρίσκει σύμφωνο. Επίσης, ε, κάνουμε ένα σχόλιο για το κοινωνικό ντάμπινγκ που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ και με αυτό. Εγώ υπέβαλα 10 τροπολογίες για αυτή την γνωμοδότηση και φυσικά απέσυρα μία τροπολογία για να μην υπάρξουν επαναλήψει. Οι συμβασίε στι οποίες φτάσαμε είναι ισορροπημένοι. Ευχαριστώ την εισηγητριά μας για την πολύ καλή δουλειά της και την ε, διάθεση συνεργασία που έδειξε. Συνεργάστηκε και με μένα και με άλλους κοιόδε εισηγητέ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ισορροπημένη έκθεση. Τίποτα άλλο. Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Φαίνεται πολύ καλά το πράγμα. Τώρα Κάποιο που ζητά τον λόγο από του ε, φιλελεύθερου. Ο Φίλιπ όμω θα παρέμβει τώρα. Έχει τον λόγο. Έχει τον λόγο, Φίλιπ. Yes. Yes, Η μία έκθεση ακολουθεί την άλλη. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της επί και για το ότι συνέταξε συμβαστικές τροπολογίες Γενικά οι απόψεις μας έχουν καλυφθεί και θα υποστηρίξουμε τις περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες. Η A και η F με βρίσκουν σύμφωνο. Η A μιλάει για το ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού για να εξασφαλίσει ισοτιμία και να επιτρέψει την ε, εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η F ε, θέλει ε, ευκρίνεια στους ε, κανόνες περί επενδύσεων, ειδικά στις κοινωνικές και οικονομικές υπηρεσίες. Η ευκρίνεια εδώ, η σαφήνεια θα ήταν πολύ καλή για όλους τους ενδιαφερόμενους. Γενικά στηρίζουμε τις ιδέες της αναβάθμισης για να μειώσουμε την ανεργία των νέων στη συμβαστική G. Ευχαριστώ που πήρατε τις απόψεις μας υπόψη. Ένας βαθμός ευελιξίας σε σχέση με όλα όσα συνεισφέρουν στο, σε ένα σωστό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μας βρίσκουν ε, σύμφωνους. Για το AIDS ε, χαιρόμαστε για την ε, επικοδομητική της πνεύμα. Ο διάλογος που έγινε από τον Επίτροπο Ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει τον δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε το ρόλο μας, ούτως ώστε η πολιτική ανταγωνισμού να ευθυγραμμίζεται με άλλες τοπικές και εθνικές προτεραιότητες. Ευχαριστώ επίσης τον Κόζα για τις ε, επικοδομητικές πρωτολογίες, περισσότερες από αυτές, ε, τις υποστηρίζω ολόθερμα. Γενικά νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ευρύ ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Φίλιπ. Υπάρχει κάποιο άλλος που δεν ήταν σκιώδης και θέλει να παρέμβει. Δεν υπάρχει κανείς, όχι. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Η κυρία Μπρόμς. Έχετε τον λόγο. Ε, δεν είναι εδώ η κυρία Μπρόνς και δεν έχουμε σχόλια σε αυτή τη φάση. Έχετε σχόλια. Πολύ καλά. Και τώρα εσύ, Φρανσουάς. η σειρά σου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Τους τους ευχαριστώ και εγώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τη στάση τους που ήταν πολύ επικοδομητική και συνεργάσιμη. Είναι καλή το κείμενό μας και ελπίζω η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων τη λάβει υπόψη. Ευχαριστούμε Φρανσουάζ. Αύριο θα ψηφίσουμε λοιπόν και η ΕΚΟΝ θα το κάνει αυτό στις 17 Οκτωβρίου. Επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Η κυρία Παπαδοπούλου έχει τον λόγο. Αντιγόνη Παπαδοπούλου βρίσκεται καθοδόν όμως προς τα εδώ. Να περιμένουμε δύο λεπτά να φτάσει. Τι λέτε εντάξει. Okay. Ε? Εντάξει. Για δύο λεπτά θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Εντάξει ευχαριστώ. Λοιπόν κυρίε και κύριοι μπορούμε να συνεχίσουμε. <clears throat> Μια και είμαστε στο διαδίκτυο, εκατοντάδε χιλιάδε Ευρωπαίοι μας παρακολουθούν, να επεξηγήσω για άλλη μια φορά. <clears throat> Τηρούμε πάντα την ημερήσια διαταξή μα ω ήθιστε. Πολλοί ευρωβουλευτέ που προσέρχονται όμω εδώ είναι ταυτόχρονα μέλη σε άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Πρέπει να είναι και εκεί παρόντε, προετοιμάζονται ψηφοφορίε. Δεν είναι απλό το σύστημα το οποίο λειτουργεί εδώ στην Ευρωβουλή. Δεν είναι λοιπόν απουσία σεβασμού από κάποιου ευρωβουλευτέ που βρίσκονται αλλού. Πρέπει να δείξουν κατανόηση οι πολίτε μπορούμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία να πούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται με τους σωστούς ανθρώπους που εκλέγουν οι πολίτες. Για δείτε μας, είμαστε διάφανοι και σας το αποδεικνύουμε. Έχουμε μια έκθεση τώρα για ένα ενδιαφέρον θέμα για τρίτους που αφορά μελέτες και έρευνα. Πρόκειται για σεμινάρια και εθελούσια, εθελοντική εργασία όσον αφορά την εργασία ΟΠΕΡ. Αντι, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξαιρετικές ικανότητες έχει για να συντάξει αυτό και να αναλάβει αυτό το θέμα Έχετε τον λόγο κυρία Παπαδοπούλου και οι σκιώδεις εισηγητές είναι παρόντες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρόμαστε για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αντιγόνη έχεις τον λόγο παρακαλώ. Thank you very much, uh, Chair. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πράγματι, υπάρχουν τόσο πολλές συνεδριάσεις, ήμουνα αλλού. Λοιπόν, έχω επικεντρωθεί στο θέμα αυτό. Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας δόθηκε πριν τις θερινές διακοπές. Μετά είχαμε τις καλοκαιρινές διακοπές για να στείλουμε τις τροπολογίες μας. Πολλές τροπολογίες. 158 και τελικά καταφέραμε να συζητήσουμε τους σκιώδεις εισηγητές και να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχανισμό προκειμένου να μπορούμε να συζητήσουμε μαζί. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε ένα συμβασμό με τις διάφορες πολιτικές ομάδες, μια που είχαμε πολλές και διαφορετικές γνωμοδοτήσεις. Πρέπει να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολλές διαφορετικές ε, κατηγορίες στην έκθεση αυτή τόσες πολλές κατηγορίες υπηκών τρίτων χωρών, μαθητές, φοιτητέ, σε μαθητεία, οπέρ κτλ. Και να ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να τα βάλουμε όλα σε μία και μόνο οδηγία που δεν είναι ούτε συνοπτική και ούτε ξεκάθαρη για το ποιε είναι οι προθέσεις. Συζητήσαμε χθε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας διευκρινίσει τις απαντήσεις που μας έδωσε την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή Αυτοαπασχόληση. Σήμερα λοιπόν είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πω ότι προσπαθούμε να πετύχουμε συμφωνία τουλάχιστον με κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, ακόμα και αν δεν καταφέρουμε με όλες τις συμβαστικές τροπολογίες να συμφωνήσουμε, κάποιες πολιτικές ομάδες θα τις υπερψηφίσουν. Στόχος μου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας χώρος ελκυστικός για επικός τρίτο χωρών και ο καλύτερος τρόπος είναι να τους αντιμετωπίζουμε δίκαια, με ίση μεταχείριση για όλες τις κατηγορίες των εργαζόμενων και να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Ευχαριστούμε τους άλλους σκιώδες συζητητέ από τις διάφορες πολιτικές ομάδες για το πνεύμα συνεργασίας, όπως επίσης και το προσωπικό της Επιτροπή μας. Από τις 20 αυτές συμβαστικέ τροπολογίες να ξέρετε ότι υπάρχουν μερικές πάνω στις οποίες θα συμφωνήσουμε, είτε με το ΑΕΛΚ, είτε με τους Πρασίνους, είτε με την ΑΛΤΕ. Προσπαθούμε τελικά να έχουμε και νέες συμβιβαστικές ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Οι τρεις κύριες κατηγορίες πάντως με τις οποίες είχαμε πρόβλημα ήταν η ηλικία. Κάποιοι είπαν από 18 με 35, ναι. άλλοι 18 με 30 για τους ΟΠΕΡ. Εγώ είπα ότι πρέπει να μπει ανώτατο όριο, γιατί η ΟΠΕΡ δεν μπορεί να είναι 40-50 χρονών. Πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Οπότε ή 18 και 30 θα είναι ή 18 και 35. Αν καταλήξουμε σε συμβιβασμό για το ανώτατο όριο, τότε θα έχει λυθεί. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν οι ώρες εργασίας των φοιτητών. Εάν από τρίτη χώρα έρχονται στις χώρες μέλη για να δουλέψουν, πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο αριθμό ωρών. 10 ώρες λέμε τουλάχιστον εδώ υπάρχουν διαφορέ. Οι πολιτικέ ομάδε το βλέπουν διαφορετικά όσον αφορά το ανώτατο όριο. Αλλά για να σα πω την αλήθεια, το κράτος μέλος πρέπει να αποφασίσει πόσοι είναι επιλέξιμοι και για πόσε ώρε η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Και το κύριο ζήτημα στο οποίο είχαμε τι μεγαλύτερε διαφορέ είναι το θέμα τη ίση μεταχείριση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε του ερευνητέ να του βάλει σε μια προνομιούχα θέση, να του επιτρέψει για παράδειγμα όταν τελειώνουν την έρευνά τους να μπορούν να μείνουν στη χώρα μέλους για 6 μήνες ή για 12 μήνες και να μπορούν και να βρουν δουλειά ή να ανοίξουν μια δικιά τους επιχείρηση. Αυτή η κατηγορία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έπρεπε να επιλεγεί για ίση μεταχείριση. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει με τις άλλες κατηγορίες, όπου πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχει ίση μεταχείριση εάν σύμφωνα με την ενία άδεια εργασίας θεωρούνται εργαζόμενοι. Αν μπορούν να δουλέψουν με την ενία αυτή άδεια, τότε θα έχουν ίση μεταχείριση. Αυτό είναι το τομέας πάνω στον οποίο συζητάμε ακόμα με τις πολιτικές ομάδες για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος συμβασμός και μετά από αυτή τη συνεδρίαση έχοντας ακούσει τι θα πούν οι άλλοι σκιώδες, θα βρεθούμε και τις νέες συμβαστικές τροπολογίες θα σας τις στείλω όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί αύριο πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ και για την βοήθεια των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ θέρμα. Ε, θα συνεχίσετε να εργάζεστε απόψε, έτσι, έχετε όρεξη. Έχετε κι εσείς όρεξη από το ΕΚ. τι λέτε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για όλες τις, τις προσπάθειες μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα χτες και σήμερα προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε έναν καλό συμβιβασμό και είμαι σίγουρη ότι θα πετύχουμε το στόχο μας πριν από αύριο και θα μπορέσουμε έτσι να ψηφίσουμε. Όπως είπε και η συγκήτρια, όταν επέκτηνε το στόχο από φοιτητέ, ερευνητέ και στις διάφορες άλλες κατηγορίες, δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Κυρίως γιατί έχουμε την οδηγία για την ενιαία άδεια και γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε την γραμμή που υπάρχει ήδη. Όταν όμως φτάνουμε στην ίση μεταχείριση πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πιο ευνοϊκή μεταχείριση στους εργαζόμενους ή γενικά στους πολίτες από τρίτες χώρες σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό οι συμβαστικές τροπολογίες F και κάποια άλλη για το άρθρο 21 και για την αιτιολογική σκέψη 36 μας δημιουργούν πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα δικαιώματα με την οδηγία αυτή. Ότι θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την οδηγία για την άδεια πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό και η διατύπωση θα ήθελα να αλλάξει λίγο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα επιτρέψουμε η ίση μεταχείριση με ε, επικόους από την ίδια τη χώρα. Πρέπει να είναι σαφής εδώ η διάκριση. Γι' αυτό θέλω να προσθεθεί μια πρόταση που να λέει ότι μόνο εάν θεωρούνται από το κράτος μέλος ως εργαζόμενοι και έχουν γίνει δεκτοί στο κράτος μέλος για να δουλέψουν θα υπάρχει αυτή η, η συμμεταχείριση. Γιατί η ενία άδεια δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να έρθει στο κράτος μέλος και να δουλέψει εκεί. Του δίνει αυτή τη δυνατότητα με μία ενιαία άδεια. Και τότε μιλάμε για εργαζόμενους. Ενώ εδώ, με αυτές τις νέες κατηγορίες, μερικές φορές είναι εργαζόμενοι, αλλά οι ΟΠΕΡ, για παράδειγμα, δεν έχουν ε, σύμβαση εργασίας. Είναι κάτι διαφορετικό. Ή όσοι ακολουθούν μαθητεία και αμείβονται. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι να έχουν μεν κοινωνική ασφάλιση, αλλά δεν είναι εργαζόμενοι. Βάσει του συστήματος ενίας άδεια όμως θα μπορούσαν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς διατυπώνουμε αυτές τις τροπολογίες. Με τους σκέφτες από τις άλλες πολιτικές ομάδες πάντως καταλήξαμε σε αρκετά καλούς συμβιβασμούς και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας πριν από αύριο το πρωί και θα είμαστε έτοιμοι αύριο. Ευχαριστώ πάλι την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχόμαστε καλή διασκεδαστική βραδιά και εσείς θέλετε να συμμετάσχετε για τους άλλους συμβιβασμούς. Τι λέτε? Yes, thank you. Well, some of us... Ευχαριστώ. Ναι, κάποιοι από εμά σήμερα το βράδυ έχουμε πολλή δουλειά. Τι να κάνουμε. Αλλά απ' την άλλη για τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε τώρα μπροστά μας. Καταλαβαίνουμε ότι είχαμε λίγο χρόνο όλοι στη διάθεσή μας. Πάντως εμείς πιστεύουμε ότι οι συμβαστικές τροπολογίες πηγαίνουν σε διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι οι τροπολογίες μας. Οπότε το όνομά μας δεν νομίζω ότι θα έπρεπε καν να βρίσκεται στις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Το ένα ζήτημα που μας απασχολεί είναι το θέμα της ίσης μεταχείρισης. Για μας, πάντα λέγαμε ότι πρέπει να έχουμε την μπλε κάρτα και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε για την ενιαία άδεια. Μπερδεύω τα λόγια μου, λέω μιλήτρια. Δεν θέλουμε να πάμε πίσω όσον αφορά τους ερευνητές και την μεταχείρισή τους. Τώρα για τον χρόνο εργασίας και ποια θα είναι η βάση, θέλουμε να δεχτούμε τις 20 ώρες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε αν κάποιοι θέλουν 10, εμείς δεν θα θέλαμε να υπάρχει ανώτατο όριο. Γιατί από την εμπειρία που έχουμε σε διάφορες χώρες μέλη, ακόμα και όταν υπάρχει ανώτατο όριο, τελικά αποτελεί στοιχείο εκφοβισμού για αυτούς που μπορεί να δουλέψουν μια-δυο ώρες παραπάνω. Ότι αν το ξεπεράσετε δηλαδή οι αρχές θα έρθουν και θα σας ζητήσουν το λόγο. Όσον αφορά την ηλικία των ΟΠΕΡ, ξέρω ότι από το 69 υπάρχουν ε, συμφωνίες. Θα έπρεπε να ευθυγραμμιστούμε με την σημερινή πραγματικότητα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι υπάρχουν πολύ επιτυχημένα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πιο μεγάλους ανθρώπους ηλικία που δουλεύουν ως ΟΠΕΡ και που δεν είχαν τη δυνατότητα όταν ήταν 18 ή που δεν ένιωθαν ότι μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά τότε. Γι' αυτό και καταθέσαμε την τροπολογία μας. Φαντάζομαι ότι ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες θα υπάρξουν συμβιβασμοί, αλλά η δικιά μας ομάδα μάλλον δεν θα συμμετάσχει, από ό,τι φαίνεται. Λυπάμαι. Εντάξει, σαφή τοποθέτηση. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλοι ευρωβουλευτέ που θέλουν να ζητήσουν λόγο, που δεν είναι σκιώδει συζητητέ. Όχι, δεν υπάρχει κανεί. Φίλιπ, όχι έτσι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θέλει να παρέμβει, αντί για την κυρία Χίος. Όχι έτσι. Όχι για αυτό το θέμα. Εντάξει, ευχαριστώ. Ο κύριος Σούιτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα περιοριστώ σε κάποια σχόλια για το θέμα το οποίο ήδη συζητήθηκε σε προηγούμενες συναντήσεις και συζητήθηκε και σήμερα ελάχιστη ίση μεταχείριση. Και να παρουσιάσω και πάλι την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθέτησε όσον αφορά τους ερευνητές. Και για να μην οπισθοδρομήσουμε όσον αφορά τα δικαιώματα ίσης μεταχείρισης των οποίων απολάβουν ε, ε, σε σχέση με τη σημερινή οδηγία χρειάζεται μια παρέκκληση, μικρή παρέκκληση από την οδηγία για την ενιαία άδεια ή αδειοδότηση. Αυτό προτείνουμε. Για τους φοιτητές τι λέμε προτείνουμε να μην εξαρτάται η δική τους δικαιοδοσία ή όχι για αυτή την ενιαία άδεια αν μπορούν να εργαστούν ή όχι πρέπει να καλύπτονται πλήρως από την ενιαία άδεια. Αυτό συμπεριλαμβάνει όμως το γεγονός ότι υπάρχουν και κάποιες πιθανές εξαιρέσεις για τα κράτη-μέλη υπό το καθεστώς της ενιαίας άδειας για τους φοιτητές. Δεν θα αμφισβητήσουμε λοιπόν αυτές τις εξαιρέσεις για τα κράτη-μέλη, για τις υπόλοιπες ομάδες. Όλοι, όλες θα πρέπει να δικαιούνται ίση μεταχείριση υπό αυτή την οδηγία, αλλά μόνο όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και και Και όπως από πλευρά εισηγητού αναφέρθηκε, εκείνοι που υπό το εθνικό δίκαιο ή το κοινοτικό δίκαιο θα θεωρούνται ότι εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούν να έχουν αυτή την κάλυψη και όχι μόνο για τις ε, υπηρεσίες και αγαθά αλλά για όλες τις άλλες περιπτώσεις υπό την ενιαία άδεια. Αυτό νομίζω αποσαφηνίζει τη θέση της Επιτροπής για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση με την Αντιγόνη. Να δούμε τι θα γίνει απόψε Αντιγόνη για αυτά τα θέματα που θα καταλήξετε. Yes, Νομίζω... Σίγουρα θα το καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε και να καταλήξουμε και σε ε, μια καλή συμφωνία. Θα βρούμε ένα συμβιβασμό σε σχέση με τις προτάσεις και των πρασίνων για ανώτατο όριο όσον αφορά τις 20 ε, ώρες για να, τους ε, να μπορούσαμε να τους ικανοποιήσουμε και θα έχουμε και μια τροπολογία για ένα θέμα το οποίο θα καταθέσω γραπτός τη διατύπωση δεν θέλουμε να είμαστε προκατηλημένοι στις θέσεις μας. Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις πολιτικές ομάδες στα αιτήματά τους με μια μέση οδό που ακολουθούμε. Και σύμφωνα με τις συζητήσεις που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εχθές, πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το οποίο μας ανέφεραν σε σχέση με το άρθρο 36 που καθορίζει ακριβώς ε, τι γίνεται σε σχέση με τους αμοιβόμενους και μη αμοιβόμενους μαθητευόμενους και εξασκούμενους ε, και να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με το άρθρο 79 της συνθήκης. Διαφορετικές κατηγορίες σε σχέση με τους φοιτητές και τις πιθανές εξαιρέσεις, πώς διαφορετικά θα μπορούσαν να υλοποιηθούν όλα αυτά, έχοντας υπόψη αυτό το έγγραφο το οποίο μας διατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω θα καταλήξουμε σε συμφωνία και αύριο θα έχουμε τον κατάλογο ψηφοφορίας έτοιμο και οι συμβιβασμοί θα είναι με όλες τις τρεις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Και εδώ σαφέστατη τοποθέτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο λοιπόν και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τον Οκτώβριο, 17 Οκτωβρίου θα ολοκληρώσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, η Edit Bauer προβλέπεται στον κατάλογο μου, αλλά περιμένουμε, τι λέτε. Είναι εδώ κοντά, θα έρθει σε λίγο, τι λέτε. Γιατί διαφορετικά προβληματίζομαι να δω αν μπορούμε την Jean Lambert να πάρουμε πιο πριν. Jean, παρίστασε, Jean Lambert, να το κάνουμε Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον. Να το κάνουμε Παρακαλώ. Συμφωνείς, έχεις τον λόγο λοιπόν. Παρακαλώ. Uh, Μαύρο το φάκελό μου. Σας παρακαλώ. Για να μην μιλήσω για λάθος θέμα. Οι βουλευτές θα θυμούνται ότι η γνωμοδότηση που ετοιμάζουμε θα αποσταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία ε, συμμετέχει στα πλαίσια της διαβούλευσης ε, που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή για το θέμα των πλαστικών. Με βοήθειά Και προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα θέματα, τα σχετικά που μπορεί να επηρεάσουν την απασχόληση. Ε, πρέπει να δούμε τις διαστάσεις της υγείας, της ασφάλειας και της κατάρτισης όμως. Είχαμε διάφορες τροπολογίες από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και γενικά νομίζω ότι όλες αυτές τις τροπολογίες, σχεδόν το μήνυμα 331, μπορώ να τις χαρακτηρίσω επικοδομητικές, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Είμαι ευγνώμων προς αυτούς και προς αυτούς τους συναδέλφους που τη συνέταξαν. Μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς, ειδικά στις παραγράφους που έχουμε πολλαπλές τροπολογίες. Παράγραφος 1 που μιλάει για θέματα αξιολόγησης, αξιολόγησης των τεχνολογιών ε, σε σχέση με το περιβάλλον. Προσπαθούμε να βρούμε ένα συμβασμό που να βασίζεται ε, στη τροπολογία του Jean-Luc Μπενάμιας, γιατί μιλάει για πολύ σημαντικά θέματα αυτή η τροπολογία. και με άλλους συναδέλφους ε, μπορούμε να ψάξουμε λίγο την ε, διατύπωση. Για την παράγραφο 2 είχαμε έξι υποβληθήσεις τροπολογίες που στηρίζουν τομείς που έχουν καλό δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για το συμβασμό μπορούμε να στραφούμε στους τρεις άξονες. Καταρχάς, να φτιάξουμε ποιοτικέ θέσει απασχόληση, να είναι αξιοπρεπή αυτή η απασχόληση δηλαδή, ε, Παραδείγματο χάρη ανακύκλωση των πλαστικών, εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση. Επίση, ε, ανάπτυξη μια οικονομία με χαμηλέ εκπομπέ διοξείδιου του άνθρακα, δεύτερο άξονα. Και τρίτο άξονα, ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών και διαφόρων φορέων. Νομίζω ότι μπορούμε να επεκταθούμε γύρω από αυτούς τους άξονες. Παράγραφος 4. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συμβασμός. Μπορούμε να αναφέρουμε τα θέματα που γίνουν τροπολογίες. Ίσως όμως η τροπολογία 19 της κυρίας Παπαδοπούλου μιλάει για κάποια νούμερα τα οποία συνδέονται με την τροπολογία 2. Επομένως, ε, θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε αυτά τα επιχειρήματα της τροπολογίας 19 και 2. Παράγραφος 5 λέει και καινοτομία στον τομέα αυτό. Νέε τεχνολογίε, πώ μπορούν να εφαρμοστούν, πώ μπορούμε να μετρήσουμε τον κίνδυνο και εδώ μπορούμε να βρούμε συμβιβασμό στην, να, για να εντάξουμε τις απολογίες 22 και 23. Οι 24 μπορούμε να τις συζητήσουμε λιγάκι, είναι πιο συζητήσιμη αλλά με μία μικρή διατύπωση νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε συμφωνία. Παράγραφος 6. Ε, δεξιότητες και κατάρτιση. Πρέπει να δούμε τα επιχειρήματα που μπαίνουν εδώ, ούτω ώστε να εντάξουμε πολλά από τα επιχειρήματα των συναδέλφων για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς όφελος κατάρτισης, για την βελτίωση του επίπεδου της εργασίας σε διάφορους τομείς. Παραδείγματο χάρη, ο τομέας της ανακύκλωσης, ε, επειδή καταγίνεται με τα σκουπίδια, αυτές τις απασχόλησεις θεωρούνται σκουπίδια. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τον κόσμο για να καταλάβει την σημασία αυτών, αυτής της δουλειάς που γίνεται για να μπορούμε να βρούμε και το, κατάλληλα, το κατάλληλο προσωπικό με τις απαραίτητες δεξιότητες. Υπάρχουν δύο-τρεις χωριστές τροπολογίες επίσης. Η μία ασχολείται με θέματα, ή μάλλον δύο, μιλάνε για θέματα εξαγωγής αποβλήτων σε διάφορες χώρες και πώς επηρεάζονται τις χώρες από αυτές τις εξαγωγές. Η μία είναι δική μου και μπορώ να τη δεχτώ βεβαίω. Αλλά και την άλλη μπορώ να δεχτώ για το θέμα τη εξαγωγή αποβλήτων και μια άλλη χωριστή τροπολογία, ε, η 16 του Ζαν Λίουκ Μπεναμία, που είναι πιο ευρεία τροπολογία και αυτή μπορώ να τη δεχτώ. Επομένω, όλε τι προτάσει μπορούμε να τι εντάξουμε και να φτάσουμε σε ένα κείμενο καλό, το οποίο θα το δεχτεί τελικά στην ε, Εκθεσής η Επιτροπή ε, Απασχόληση. Ε, Ευχαριστώ πολύ και για την προσφορά στο Σκιώδης. Η Αντιγόνη είχε, ήταν παρούσα. Τώρα παρακαλώ έχετε τον λόγο ως Σκιώδης για τους σοσιαλιστές. Έχετε τον λόγο. Μικρόφωνο. Είμαι λίγο μπερδεμένη. Γιατί διαρωτώ μου τι θα γίνει τελικά με την προηγούμενη έκθεση. Έχω να κάνω σχόλια και για αυτή την έκθεση πάντως. Μια στιγμή, να βρω εδώ πέρα τα χαρτιά μου. Σε αυτή την, σε αυτή έκθεση, ε, η Ευρωπαϊκή, ορίζοντας Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, θα πρέπει να εξασφαλίσει μια έξυπνη, βιώσιμη και με ένταξη όλων ανάπτυξη. Για δύο-τρεις τροπολόγιες έχουμε δισταγμούς. Έχουμε υπογράψει Έχουμε υπογράψει και καταθέσει περίπου 7 τροπολογίες και εστιάζουμε κυρίως στην ανάγκη του να λάβουμε υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις της νέας περιβαλλοντικής πολιτικής. Στις τροπολογίες μας αναφέρουμε ότι η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξοικονομεί 72 δισεκατομμύρια το χρόνο και μπορούμε να βρούμε και άλλα 42 εκατομμύρια, ε, δισεκατομμύρια συγγνώμη, ε, στον τομέα της ανακύκλωσης και να δημιουργήσει και πολλές θέσεις απασχόλησης. Πολύ μεγάλα τα νούμερα αυτά, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Επίσης η ανακύκλωση των πλαστικών από μόνη της ε, μπορεί να δημιουργήσει 160.000 θέσεις απασχόλησης στις 27 χώρες. Εάν αυξήσουμε το επίπεδο ανακύκλωσης μέχρι 70% μέχρι το 2020. Θέλουμε λοιπόν να υποβάλουμε τις τροπολογίες αυτές για να ε, δούμε ότι υπάρχει δυναμικό απασχόληση στο τομέα της ανακύκλωσης και δεν θα πρέπει όμως αυτό να υποσκάψει τις δυνατότητε για να μειώσουμε τη χρήση των πόρων. Γιατί και αυτή είναι μια άλλη πρόκληση και αυτή προσφέρει ε, θέσεις απασχόλησης. Γενικά, οι περισσότερες ε, τροπολογίες μας βρίσκουν σύμφωνους και μόνο δύο-τρεις μας προβληματίζουν. Ε, αυτό θα αντικατοπτριστεί στην αρνητική ψηφοφορία μας, στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους ε, φιλελεύθερους ο Φίλιπ και πάλι. Συνεχίστε Φίλιπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά ήμουν σκιώδης συζητητής για αυτή την έκθεση, γιατί επί πολλά χρόνια απασχολούσαν ε, και συχαινόμουν τα πλαστικά απόβλητα. Επομένω, μεγάλη χαρά συμμετείχα στη δουλειά. Συμφωνώ με την εισηγήτρια για τη διαχείριση των αποβλήτων, ειδικά των πλαστικών αποβλήτων και η οικολογική καινοτομία έχει σοβαρό δυναμικό για να δώσει νέες θέσεις απασχόληση σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι θα πρέπει οι πολίτες να έχουν τι απαραίτητε ε, δεξιότητες για να έχουν πρόσβαση απασχόληση. Και επίση το στάτου των θέσεων αυτών στην ε, βιομηχανία αποβλήτων πρέπει να βαθμιστεί. Ε, επίσης ε, είδατε την διαφορετική σημειολογική, τη, σημειολογική σημασία του όρου απόβλητα, ανακύκλωση, διαχείριση μάλλον αποβλήτων, έχει σημασία του αυτό. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε για τα ωφέλη της επαγγελματικής κατάρτισης και της διαβίου μάθησης και έχω υποβάλει τροπολογία. Η πλειοψηφία των τροπολογιών είναι θετική και θα μπορέσουμε να υποστήριξουμε τις περισσότερες τροπολογίες. Περιμένω τη συνεργασία με τους υπόλοιπους κοιόδης εισηγητές και με την εισηγήτρια για να υποβάλουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Σε ευχαριστώ θερμά, Φίλιπ. Κάποιος ευρωβουλευτής που θέλει να παρέμβει ακόμη, αλλά δεν είναι σκιώδης, παρακαλώ. Δεν υπάρχει κανεί. Ωραία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Η κυρία Στέφνερ παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Συγγνώμη, Frau δεν παρίσταται κυρία Στέφνερ. Δεν έχουμε σχόλια λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συντομεύουμε λοιπόν έτσι. Τζιν, έχετε τον λόγο. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια λεπτά παραπάνω, αν θέλετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνήθως ένα-δύο λεπτά μας δίνουν όταν έχουμε παραπάνω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα τόσο χρήσιμα σχόλιά σας. Συμφωνώ ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν αναρωτιόμαστε πού θα βρούμε νέες θέσεις απασχόλησης. Να, ένα τομέα ο οποίος μπορεί να προσφέρει θέσεις απασχόλησης. Σίγουρα βέβαια τα θέματα για την επαγγελματική κατάρτιση έχουν πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Και άλλα πράγματα που είπαν οι συνάδελφοι, κατά πόσο εμπίπτει στο θέμα της μείωσης της εξάρτησης των πόρων 50% των πλαστικών καταλήγουν στις χωματερές σήμερα και δεν χρησιμεύουν για τίποτα σε ολόκληρο τον πλανήτη, ούτε βέβαια και για την οικονομία, ούτε για την απασχόληση. Άρα εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ξέρω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος επίσης το εξετάζει από τη δικιά της οπτική γωνία, για το θέμα δηλαδή των πόρων. Για να μην καταλήγουν στους ωκεανούς, στις χωματερές και να δημιουργούν άλλα προβλήματα. Άρα ναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι χρήσιμο με αυτό. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Θα βρεθούμε για τους συμβασμούς. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και για την προθυμία να δείξετε ελαστικότητα για το χρονοδιάγραμμα. 17 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε και η Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 5 Νοεμβρίου θα ψηφίσει προς έγκριση και ελπίζουμε ότι θα δεχτεί όλες τις έξυπνε ευφυείς σκέψεις μας. Αγαπητή Edith Bauer, Τώρα έχεις εσύ τη σειρά να παρέμβεις. Θα θέλαμε να καλύψουμε την καθυστέρηση. Το σημείο σου χρειάστηκε να το πηδήξουμε για να περάσουμε σε επόμενο, επειδή ήσουν σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Η διάσταση του φίλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρωμά, των Τσιγκάνων. Αυτό είναι το θέμα σου. Έχεις τον λόγο, Edith Bauer. Παρακαλώ. you uh, το είδατε. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το τελευταίο λεπτό προσπαθούσα να βρω κάποιους ε, λογικούς συμβιβασμούς και ανταλλάξαμε απόψεις ακριβώς και μόλις για κάποια από αυτά τα θέματα. Δέκα συμβιβασμούς έχουμε. Οι πιο πολλοί από αυτούς τους συμβιβασμούς υποστηρίζονται <clears throat> από ένα μεγάλο τμήμα πλειοψηφία των ομάδων Υπάρχουν όμως και κάποια, κάποιες παρανοήσεις ακόμα για ένα θέμα για την απασχολησιμότητα για παράδειγμα κάποιων ατόμων. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και ακαθόδες. Όμως είμαι βεβαία ότι η απασχολησιμότητα και η θετική απασχολησιμότητα, δυνατότητα απασχόλησης σε συνδυασμό με το μεγάλο, τη μεγάλη ομάδα των Ρωμά που παραμένουν χωρίς εκπαίδευση και εγκαταλείπουν το σχολείο είναι ένας από τους λόγους επίσης πέρα από την αρνητική διακριτική μεταχείριση, πέρα από την έλλειψη ε, θέσεων εργασίας και απασχόλησης, πέρα από την δυσκολία απασχολησιμότητας πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουμε τα μάτια και να αγνοήσουμε το ότι υπάρχει πολύ χαμηλό ποσοστό ισχνή απασχολησιμότητα για τους Ρωμά, για τους Τσιγκάνους. Όσον αφορά τον συμβιβασμό Β, έγινε η προσπάθεια να εξευρεθεί κάποια λύση και είχα την εντύπωση ότι και κάποιοι συμβιβασμοί θα μπορούσαν κατά τα άλλα να είναι αποδεκτοί επίσης. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούγεται. Πίστευα ότι θα ήμουν η επόμενη εγώ, λέει η κυρία Γκέντς. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία με την Edith Μπάουερ για αυτό το θέμα ήταν πολύ θετική. Την ευχαριστούμε. Είχαμε διάφορες συζητήσεις βέβαια για κάποια θέματα, αλλά όπως επίσης και το αναφέρατε, το πώς θα διατυπώσουμε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Περισσότερο με έναν τρόπο που θα τονίζει τον ατομικό χαρακτήρα και τις ατομικές ε, ιδιομορφίες αυτού του προβλήματος ή οθετώντα μια πιο γενική συστημική προσέγγιση που θα συσχετίζεται με όλα αυτά τα πολύ περίπλοκα και σύνθετα θέματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα της κοινότητας ε, των τσιγκάνων, των Ρωμά, ακόμα και των γυναικών τσιγκάνων που ζουν ε, αποκλεισμένες ε, και στο περιθώριο και υπάρχουν προβλήματα για τη σχολική εκπαίδευση και δεν υπάρχει πρόσβαση και προσπελασιμότητα σε απασχόληση, ευκαιρίες απασχόλησης κτλ. Ήταν πολύ καρπερή, η συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Και για να τονίσουμε αυτό και να δούμε αυτές τις πτυχές που είναι σημαντικές και που δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τα διαρθρωτικά προβλήματα. Η Εντίτα υποστήριζε την άλλη προσέγγιση. Έχουμε ακόμα μια συμβαστική τροπολογία διότι διστάζουμε να πούμε αν μπορεί η σοσιαλδημοκρατική ομάδα να υποστηρίξει όχι. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που θα μπορούσε να ήταν αποδεκτή από όλους. Η παράγραφος αυτή είναι η συμβιβαστική τροπολογία ΑΒ ή ΒΑ, ΒΑ όπου για το πρώτο τμήμα κάνουμε λόγο για τα θέματα της ε, <clears throat> εγκυμοσύνης ε, των νέων κοριτσιών. Early, ε, και αν η συνειδητοποίηση των προβλημάτων σε σχέση με τον πολιτισμό των Ρωμά μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Και πάλι, εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Δεν είναι πολιτισμικό χαρακτηριστικό της κοινότητας των Ρωμά. Είναι περισσότερο επίπτωση αποτέλεσμα μιας απελπιστικής κατάστασης ακόμα και η ε, εκπαίδευση δεν μπορεί να οδηγήσει στην απασχόληση. Και το αμόνα έσοδα θα μπορούσαν να είναι τα επιδόματα πολυτεχνίας που βασίζονται στον αριθμό των παιδιών που έχουν αυτές οι γυναίκες. Και ο μόνος τρόπος για να βρουν δυνατότητα διασφάλισης εσόδων για αυτή την κοινότητα, για αυτές τις νέες γυναίκες είναι αυτό και προσπαθούμε να βρούμε μια δυνατότητα γιατί με αυτή τη διατύπωση δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την τροφολογία αυτή. Δεν είναι πολιτισμικό χαρακτηριστικό των συγκάνων αυτό, των Ρώμα. Είναι χαρακτηριστικό και επίπτωση, είναι αποτέλεσμα του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης στην οποία ζουν. Αυτή είναι η συζήτηση την οποία είχαμε αναπτύξει και είχαμε όλο το χρονικό διάστημα για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια λύση που θα ήταν αποδεκτή. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε θερμά Κίνγκα και για τις πολλές πληροφορίες που μας έδωσες. Και πάλι ο Φίλι Μπένιον παρακαλώ τώρα. Έχεις τον λόγο Φίλι. Μέρος uh, του κύριου Κατσίν. Λυπάται δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μας. Συζήτησα όμως το θέμα και δεν θα διαβάσω απλώ το σημειωμά του, αλλά θα σα διαμηνήσω τα σχόλιά του. Ε, καλωσορίζουμε την έκθεση τη πρωτοβουλία και την ε, γνωμοδότηση τη πρωτο... Επιτροπής. Υπάρχουν λίγες ε, τροπολογίε που δεν μπορούμε να στηρίξουμε, γιατί θα μπορούσαν να σημαίνουν ω ως ε, στιγμάτιση των α, γυναικών Ρωμά. Βασικά είναι οι ίδιε επιφυλάξει με της κυρίας Κίνγκα. Πρέπει να διατηρήσουμε και ένα βαθμό πολιτικά ορθούς όλη αυτή την ιστορία. Είναι δική μας ε, γνωμοδότηση, ίδιας πρωτοβουλία, είναι ευαίσθητο το θέμα και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν δεν θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιλύουν. Γι' αυτό λοιπόν ε, όταν μιλάμε για τη σεξουαλική εκπαίδευση, πρόορη εγκυμοσύνη, υψηλά ποσοστά εγκατάσταση του σχολείου, χαμηλά ποσοστά απασχολησιμότητας. Ε, αυτά είναι απλουστευτικά και στιγματίζουν ε, ομάδες. Αυτό τον όρο, ειδική ε, εθνική ή εθνοτική ομάδα, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. γιατί μπορεί να σημαίνει και ειδικά κοινωνικά δικαιώματα. βασικά πρέπει να αλλάξουμε απλώς τη διατύπωση, την, τη φρασιολογία αυτές τις έννοιες για να μην δημιουργούν προβλήματα στην ερμηνεία. Από την άλλη, μπορούμε να υποστηρίξουμε τις περισσότερες συμβαστικέ τροπολογίε και όλες τις τροπολογίε που ε, εμπλουτίζουν το κείμενο. Γενικά υπάρχει συνένεση, συμφωνούμε με τις λύσεις και δεχόμαστε γενικά την ε, σύγκληση αυτή που υπάρχει. Πρόεδρος, δεν έχω άλλο ευρωβουλευτή στον κατάλογο μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα λοιπόν. Η κυρία Τσίνη, έχετε τον λόγο, εντάξει. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η θέση της Επιτροπής όσον αφορά τις γυναίκες Ρώμα είναι από το 2011 ότι αυτές υποφέρουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό και από τις διακρίσεις. Και αυτό βέβαια φαίνεται στη γνωμοδότηση της εισηγήτριας. Στην τέταρτη διεθνή διάσκεψη για τις γυναίκες Ρώμα, όπου συμμετείχε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, οι γυναίκες Ρωμά αναφέρθηκαν σε πολλά ευαίσθητα ζητήματα. Η συζήτηση που γίνεται εδώ και αναφέρεται στα πολιτιστικά ή άλλα ζητήματα άπτονται δικαιωμάτων των γυναικών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολλές φορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται λοιπόν το ζήτημα και υπενθυμίζει ότι πράγματι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε για να μην στέλνουμε ένα μήνυμα το οποίο κινδυνεύει να παρεξηγηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η συγγήτρια θα έχει τον τελευταίο λόγο, η κυρία Έντιτ Μπάουερ. Θα ψηφίσουμε αύριο. Λοιπόν, ποια είναι η θέση σου, Έντιτ. Ευχαριστώ. Κοιτάω τις τροπολογίες. Νομίζω ότι η τροπολογία 20, η οποία μιλάει για αυτές τις πολιτιστικές πτυχές, βγαίνει από το πακέτο. Και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση ερμηνείας όπως αυτή που αναφέρατε. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω, κύριε Πένιον, ότι δεν σκοπεύουμε να στεγματίσουμε ούτε προθέσει έχουμε να στιγματίσουμε οποιονδήποτε. Προσπαθούμε να μιλήσουμε για θέματα απασχόληση. Είναι και θέμα αρμοδιότητάς μας. Και να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό απασχόληση των Ρωμά. Ποιο είναι ο λόγος. Η Κίνκα Γκάντ έχει απόλυτο δίκιο. Είναι περίπλοκο το θέμα. Και δεν θέλουμε μονοκόμματες απόψεις μονοδιάστατες. Φυσικά, το λάθος δεν είναι μόνο των ατόμων. Αυτοί φταίνε που είναι φτωχοί. Από την άλλη, ούτε οι κοινωνίες ήταν αποκλειστικά αυτές. Η κατάσταση μάλλον είναι πολύ πιο περίπλοκη. Και πρέπει να βρούμε μια λύση για αυτά τα θέματα, να βρούμε απαντήσεις. Γιατί αυτά τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ θερμά, Αύριο θα ψηφίσουμε και η Επιτροπή Γυναικών στις 14 Οκτωβρίου θα ψηφίσει για να εγκρίνει και να συμπεριλάβει πολλά από αυτά που θα έχουμε προτείνει εμείς ελπίζουμε. Ευχαριστώ θερμά. Αυτό ήταν το 11, το 12 το είχαμε, αλλά έχουμε τώρα και το 6 ακόμα που όπως θυμόσαστε πρέπει να καλύψουμε. Φίλιπ Μπουλάν, τώρα έχεις εσύ η σειρά να παρέμβεις. Πρόκειται για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της αηφορίας ε, για το θέμα της επανοβιομηχανοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σειρά να παρέμβεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε με ρωτήσανε αν μπορούσα να καθυστερήσω μέχρι να έρθει ο Φρεντερικ Ντάλενς, αλλά δεν το βλέπω να έχει έρθει. Α, είναι στο κτίριο. Καλά. Ε, θα αρχίσω με το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε ήδη για την έκθεση αυτή. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν το γενικό προσανατολισμό της έκθεσης. Είναι γνωστός. Α, να Λοιπόν, 43 τροπολογίες υποβλήθηκαν, κυρίως από τους σοσιαλιστές και τους πράσινους. Εγώ υπέβαλα τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες, οι οποίες καλύπτουν 17 τροπολογίες. Αυτές οι τέσσερις συμβαστικές στηρίζονται από τους σοσιαλιστές και από τους πράσινους και χθε το βράδυ είχαμε και κάποιες προτάσεις τροποποίησης αυτών των συμβαστικών τροπολογιών από τους φιλελεύθερους, οι οποίοι προτείνουν, όπως σας είπα, κάποιες τροποποίησεις. Αν λοιπόν συμφωνούμε με τους σοσιαλιστές και τους πράσινους τελικά να δεχτούμε τις τροποποίησεις αυτές, ευχαρίστως να πάρουμε μαζί μας και τους φιλελεύθερους. Όμως για τη συμβαστική, αριθμός, ε, τη α που προτείνεται από τους φιλελεύθερους να ακολουθήσουμε την εξής διατύπωση. Ένα κοινωνικό ισχυρό διάλογο και να προσθέσουμε και ή μια ενεργό πολιτική για την απασχόληση. Εγώ Προσωπικά θα αφήσω τον Φρεντερίκ Νταρντά να πει τη γνώμη του, αλλά δεν είμαι κατά. Δεν βλέπω γιατί να μην συμπεριλάβουμε αυτή την τροποποίηση που μας ζητάνε. Στη συμβαστική Β προτείνεται να μιλήσουμε για ατομικά δικαιώματα ε, πρόσβαση σε επιπλέον κατάρτιση. Αυτό θέλουν οι φιλελεύθεροι να προσθέσουμε και να μιλάει για το ατομικό δικαίωμα συμπλήρωσης της κατάρτισης. Αν ε, λοιπόν μας εξηγήσουν ποια είναι η διαφορά, εντάξει. Τρίτη συμβαστική τροπολογία έχει να κάνει με την ευελιξία ασφάλεια. Γι' αυτό το σημείο, αντίθετα, νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσουμε να αναπτυχθεί η ευελιξία ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο, από μόνη της τα λέει όλα. Άρα δεν θα συμφωνούσα με μια τροποποίηση αυτής της εμβαστικής τροπολογίας. Συνοψίζοντας λοιπόν, λέω, τροποποίηση, ναι, αν ο αρχικός μας συνασπισμός συμφωνεί με την Α και Β, με την τροποποίηση δηλαδή των Α και Β, ευχαρίστω. Στον κατάλογο ψηφοφορίας πάντως, εγώ θα πω να ψηφίσουμε κατά των τροπολογιών 1, 3, 9 20 και 25 που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβαστικές. Ό,τι λεπτομέρειες θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Πάντως αυτά για να συνοψίσω ότι η έκθεση αυτή δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα κατά τα άλλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Φιλιππό. Φρεντερίκ, έχεις πολλά σχόλια. Ε? Λοιπόν, σε ακούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συγγνώμη, συγγνώμη που καθυστέρησα, σχεδόν καθυστέρησα. Άκουσα όμως τα ουσιαστικά. Λοιπόν, με, με ικανοποιεί το αποτέλεσμα που έχουμε μέχρι τώρα με τον εισηγητή πώς συμπεριλήφθηκαν οι τροπολογίες μας στις συμβαστικές. Κάποια ζητήματα τα θεωρούσα πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα στόχος των επενδύσεων που πρέπει να είναι η δημιουργία και η διατήρηση της απασχόλησης, να βελτιωθεί το δικαίωμα στην κατάρτιση, στη γνώση. Ε, επενθυμίζουμε ότι οι προσπάθειες δεν πρέπει να έχουν να κάνουν μόνο με τις βιομηχανίες υψηλής προσθέμενης αξίας αλλά και με τις άλλες ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία ασφάλεια, την κοινωνική προστασία δηλαδή και την ελαστικότητα. Ε, να αναφέρεται ένας ισχυρός κοινωνικός διάλογος, η μνήμα που γίνεται στην έκθεση με αυτά που είπε ο συνάδελφος Αλεχάνδρο και να χρησιμοποιείται καλύτερα η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα των εργαζομένων. Όλα αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τώρα στις συμβαστικές τροπολογίες και χαίρομαι γι' αυτό. Έχω να κάνω όμως κάποιες παρατηρήσεις για αυτά που ζητάνε κάπως αργά θα έλεγα οι συνάδελφοι. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 1 με εκπλήσει η διατύπωση που θέλουν το και και το ή διαζευτικό. Εγώ νομίζω ότι το και ανταποκρίνεται καλύτερα στις προθέσεις μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την άμβλυνση και από το και να περάσουμε στο και ή διαζευτικό. Να τα βάλουμε και τα δύο. Συμβαστική β. το δικαίωμα πρόσβασης αντί για δικαίωμα. Εδώ νομίζω ότι από πίσω υπάρχει κάποια αποδυνάμωση του δικαιώματος πρόσβασης. Πώς, με τι τίμημα. Δεν βλέπω γιατί. Είναι δύσκολο να πω ότι είμαι υπέρ. Όσον αφορά τώρα τη συμβαστική τροπολογία γάμα, Καταλαβαίνω γιατί δεν συμφωνεί ο εισηγητής. Αυτά είναι τα σχόλια που είχα να κάνω για αυτές τις τροποποίησεις που μας φτάσαν την τελευταία στιγμή. Κατά τα άλλα είναι καλή έκθεση. Καλή έκθεση. Ωραία. Φιλίπ Καλή έκθεση. Φίλιπ, όπως πάντα εσύ για τους φιλελεύθερους, έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Συμφωνώ και εγώ ότι γενικά είναι μια πολύ καλή έκθεση. Οι τροποποίησει που ζητήσαμε είναι ελέσσονο σημασίας, αλλά μπορεί να έχουν σημαντικέ συνέπειε. Και δεν είναι τόσο ότι το ζητάμε αργά και νωρίτερα το ζητήσαμε. Αλλά δεν ελήφθη υπόψη το πόσο σημαντικό ήταν για μας. Τώρα, γιατί θέλουμε να μην βάλουμε και, αλλά να βάλουμε και ή ή σκέτο ή στη συμβαστική α. Δεν είναι τόσο θέμα πλειοψηφίας για τον κοινωνικό διάλογο. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι οι Γερμανοί συνάδελφοι έχουν πολύ ισχυρό κοινωνικό διάλογο και οι Γάλλοι. Ε, στο Βασίλειο δεν έχουμε. Και δεν νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα. Πάντως, αν δούμε ποιος τα καταφέρνει καλύτερα και ε, αντιμετωπίζει καλύτερα την ανεργία είναι η Γερμανία που έχει ισχυρό κοινωνικό διάλογο. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει μεν ισχυρό κοινωνικό διάλογο, έχει όμως ιδιαίτερα ισχυρές πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας. Γι' αυτό νομίζω ότι και οι δύο περιπτώσεις είναι θετικές. Και κοιτώντας τα γεγονότα, έχουμε 7,1% στον Ηνωμένο Βασίλειο, με μια ιδιαίτερα ενεργό πολιτική καταπολόμηση της ενεργείας, ίσως την καλύτερη σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερο ορθό να πούμε ότι μπορεί να είναι συνδυασμός ή μπορεί να είναι ή το ένα ή το άλλο. Γι' αυτό θέλω εγώ να βάλουμε και το και και το διαζευτικό ή γιατί έτσι λέμε ότι κάποιοι από εμά βρίσκουμε άλλους τρόπους να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με μια πολύ καλή πολιτική απασχόλησης. Δεύτερον, δεν ξέρω τι γίνεται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στα αγγλικά δεν το βλέπω. Εγώ βλέπετε δεν ξέρω γαλλικά, αλλά το προσωπικό μου μου λέει ότι στα γαλλικά υπάρχει, δεν υπάρχει στα αγγλικά. Εδώ θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε. Τώρα για την συμβαστική βήτα στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ντερντέν. Και πάλι, ναι, έχετε δίκιο για το δικαίωμα πρόσβασης στην διαβίου κατάρτιση. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το δικαίωμα απλώ. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μας απασχόλησε και μας. Υπάρχουν πολλά προγράμματα χρειάζεται ανταγωνισμό για να μπει κανεί. Κάνει κανεί αίτηση και υπάρχουν πολύ περισσότερες αιτήσει από τις θέσεις που τελικά είναι διαθέσιμες. Οπότε όταν κάποιος δεν μπορέσει, κάνει αίτηση δηλαδή, αλλά δεν πάρει αυτή τη θέση, τότε τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πει ότι μου το αρνηθήκανε, μα μπορεί να απέτυχε στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να πάρει αυτή τη θέση. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος παρόλο που απέτυχε στις εισαγωγικές κατά κάποιο τρόπο να επιμείνει ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης. Δεν είναι ένα απόλυτο δικαίωμα αυτό. Αυτό θέλω να πω. Σκεφτούμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η διατύπωση αυτή νομικά, γιατί όταν μιλάμε για δικαίωμα κατοχυρώνεται νομικά, έτσι. Οπότε να ξέρουμε ποιε θα είναι οι συνέπειες αν το βάλουμε. Γι' αυτό και εγώ προτιμώ να λέμε δικαίωμα πρόσβασης παρά να μιλάμε για ένα απόλυτο δικαίωμα. Τέλος, για την ευελιξία ασφάλεια. υπάρχουν δύο διαφορετικές διατυπώσεις, αλλά το ίδιο πράγμα φαντάζομαι σημαίνει έτσι, μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε κι εσείς. Μεγάλη ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά μπορούμε να μάθουμε ένα από τον άλλον. Και από την ίσο, δηλαδή από τη Βρετανία. Εντάξει, καλή ευκαιρία θα ήταν αυτή. Μετά του Σκιώδη τώρα έχουμε <clears throat> την Τανούτα, πλήρες μέλος που θέλει να παρέμβει. Έχει τον λόγο, Τανούτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα δύο φορές να παρέμβω. Πρώτη φορά εξ ονόματος του συναδέλφου Κοσουόφσκι που βρίσκεται καθοδόν προς την Ευρωβουλή και δεν το κατάφερε να φτάσει έγκαιρα. Και μου ζήτησε εγώ να παρέμβω εξ ονόματος του. Μπορώ να παρέμβω. Πολύ ωραία. Μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του συναδέλφου λοιπόν κυρίου Κοσουόφσκι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπουλόν για το έργο που επετέλεσε σε σχέση με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Το καλωσορίζω ιδιαίτερα. Είναι καλοδεχούμενο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να καταλήξουμε σε δημιουργία ενός θετικού περίγυρου για τις ε, επενδύσεις, μιας ε, θετικής ατμόσφαιρας. Να υπάρξουν ευκαιρίες και πάλι, ώστε να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε και να σημειώσουμε μια ανάπτυξη οικονομική. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένας θετικός στόχος ένας φιλόδοξος και ευκταίος στόχος. Η βιομηχανία να μπορέσει να έχει ένα ποσοστό 20% που θα διασφαλίσει σε σχέση με αυτό. Όμως να σκεπτόμαστε ότι και οι διαδικασίες βιομηχανοποίησης σήμερα είναι διαφορετικές από ό,τι στο παρελθόν σήμερα δεν έχει τόσο κέρια σημασία όπως παλαιότερα. Οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις όλο και μεγαλύτερο ρόλο διαδραματίζουν σήμερα και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τονίζεται ως στόχος, ως έργο και τονίζεται ότι πρέπει να έχουν καλύτερη διευκολυμένη προσπελασιμότητα σε υποστήριξη, κονδύλια, δάνεια, πιστώσεις. Υποστηρίζει λοιπόν με συμβουλευτικό έργο η Ευρωπαϊκή Ένωση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καλύτερες δυνατότητες, βελτιωμένες δυνατότητες για τη χρηματοδότησή τους, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην ενιαία κοινή αγορά. Εκείνο όμως το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ένα φιλικό κλίμα, ένα θετικό περίγυρος. Η άρση, η κατάργηση των προσκομμάτων και των εμποδίων για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν συμφωνώ με τις τροπολογίες 30, 28, συγγνώμη, 28 και 30. Δεν συμφωνώ με αυτές όπου πρόκειται για κατάργηση ε, φορολογικών προσκομμάτων ή επιβαρύνσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ένα μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης και πρέπει να εκπονήσουμε τέτοιες προτάσεις για να εξευρεθούν λύσεις ώστε στις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις να διευκολύνουν τη λειτουργία τους και όχι να την επιβαρύνουν, ώστε να είναι πιο εύκολο να δημιουργηθούν και νέες επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω σε σχέση με την πρώτη παρέμβαση. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο θέμα. Συμφωνώ, πρέπει να πω, με τον συνάδελφο, κυρίως με το τελευταίο τμήμα της παρέμβασής του στην εισήγησή του. Δεν κατανοώ, δεν μπορώ να κατανοήσω πραγματικά γιατί οι συνάδελφοί μας από την ομάδα των σοσιαλιστών εδώ αυτές τις διατάξεις για την κατάργηση των φορολογικών, των φορολογικών βαρών και προσκομμάτων ε, δημιουργούν τριβές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγούν, δημιουργούν περισσότερο από 90% των θέσεων ε, εργασίας στην απασχόληση. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η πτυχή λοιπόν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το δυνατόν να είναι πολυάριθμες ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχίσουν να δημιουργούν απασχόληση. Στην δική μας χώρα, για παράδειγμα, η ανεργία είναι πολύ μεγάλη έχει διονγκωθεί και γι' αυτό είναι τόσο μεγαλύτερο να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες μας, κυρίως για τους νέους μας. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή πορεία, η ορθή πορεία που πρέπει να πορευτούμε. Πρέπει να καταργηθούν τα εμπόδια, να αρθούν τα εμπόδια και προσκόμματα και να πορευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα είναι το ευκταίο. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Τελευταίος αγορητής ο Αλεχάνδρο Θέρκας. Παρακαλώ, Έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να στηρίξω κι εγώ με κάθε τρόπο τα επιχειρήματα των σοσιαλιστών από στόματος του σκιώδους εισηγητού μας, Νταρτέν. Δεν είναι αθώα όλα αυτά, το και ή δεν είναι αθώο. Άλλη η μία άποψη και άλλη η άλλη άποψη. Εμείς πρέπει να διαλέξουμε ή για τον κοινωνικό διάλογο λέτε ή για ένα κοινωνικό κράτος. Δεν συμφωνώ ότι είναι ή το ένα ή το άλλο. Και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το επιχείρημα αυτό του κ. ότι το Ηνωμένο Βασίλειο το είπε. Από όσο ξέρω, δεν ε, συμπεριλαμβάνεται στο πρωτόκολλο 14 του Μάστριχτ. Δεν θέλαν να συμπεριληφθούν σε αυτό το κοινωνικό πρωτόκολλο. Το Άμστερνταμ όμως το εγκρίνανε και τη συνθήκη της Λισαβόνας που λέει ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί ένα κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να πούμε ή θα έχουμε ή δεν θα έχουμε κοινωνικό διάλογο. Δεν μπορεί αυτό να το διαλέγουμε. Κανείς ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί έχει δεσμευτεί πολιτικά. Ό,τι ιδεολογία και να έχει κανείς, το έχουν υπογράψει και άρα πρέπει να το τηρήσουν. Οπότε, Ο πειρασμό στον οποίο θέλει να μας βάλει ο Βρετανός συνάδελφος δεν ισχύει. Εδώ είμαστε για να είμαστε Ευρωπαίοι και όχι για να γίνουμε όλοι Βρετανοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο ευρωπαϊκός διάλογος λοιπόν είναι μια θετική εμπειρία σε πολλές χώρες. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Η κυρία... Ο κύριος Γκρούνπαρ παρακαλώ. Έχει τον λόγο κύριε. Παρακαλώ. Yes, thank you. Thank you for letting me comment and thank... Ευχαριστώ για τα σχόλια, ευχαριστώ για την γνωμοδότηση αυτή. Ακούσαμε ποια είναι τα κύρια σημεία, ένας από τους τέσσερις πυλώνες της ανακοίνωσής μας για την κατάρτιση. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι στις οικονομίες μας δεν έχουμε τις ίδιες αναμίες στα ίδια επαγγέλματα. Ξέρουμε ότι χρειάζονται περισσότεροι επιστήμονες, περισσότεροι μηχανικοί από ότι άλλα επαγγέλματα. Και αυτό προσπαθούμε να το λάβουμε υπόψη μας στις πολιτικές μας όπου εξετάζουμε ειδικού τομεί να δούμε τι προσόντα χρειάζονται εκεί και πώς μπορούμε να προκαταλάβουμε τα πράγματα και να συμπεριλάβουμε την κατάλληλη εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Έπειτα το θέμα της κοινωνικής ευθύνης. Αυτό είναι ένα άλλος τομής για τον οποίο πρέπει να ξέρετε ότι δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχε ανακοίνωση πριν μερικά χρόνια, πρόγραμμα δράσης για τη βελτίωση της κατάρτισης όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη που περιλαμβάνει και τον κοινωνικό διάλογο. πρόσβαση στη χρηματοδότηση επίση αναφέρεται στη γνωμοδότηση ένας άλλος πυλώνας. Πιστεύω ότι ευθυγραμμιζόμαστε κάλλιστα με τα όσα αναφέρει η γνωμοδότησή σας. ευχαριστούμε πολύ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να ολοκληρώσουμε, εσείς Φιλίπ, εσείς Φιλίπ έχετε τον λόγο μετά την Επιτροπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους Κιώδης και τους βουλευτές που πήραν τον λόγο για το συμβασμό 1. Μετά από αυτές τις εξηγήσει και των φιλελεύθερων, συντάσσουμε απόλυτα με την ε, γνώμη του κυρίου Θέρκας και του κυρίου Νταρντέν. Ούτως ή άλλως και εγώ είχα προτείνει να καταψηφίσουμε την ε, τροπολογία 1 του Μπάνιον, ε, που μου φαίνονταν απαράδεκτη για αυτή την έκθεση για τον κοινωνικό διάλογο. Θέλω να διατηρήσουμε το συμβασμό Α ως έχει, για τον, τον A δηλαδή. Για τον B, ε, η προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν δημιουργεί κανένα κίνδυνο. Προτείνω να το κρατήσουμε το συμβασμό ως έχει. Και για το C, κατά, ήμουν κατά της τροποποίησής του. Κρατάω και εμένα σε αυτή τη θέση. Φίλιπ Μπάνιον, θα να πω ότι το Flex Security ή Flex Security σημαίνει ακριβώς το ίδιο σε όλες τις γλώσσες μας. Ευχαριστώ την Τανούτα που ως εκπρόσωπος και εκφράζοντας προσωπική της γνώμη ε, μίλησε για την θετική στάση που πρέπει να έχουμε στην Ευρώπη απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ευχαριστώ. Η τροπολογία 30 όπως 28 και 29, ε, την οποία δεν είχα αναφέρει, ε, δεν τη συμβρίσκω, δεν την συμμερίζομαι. 1, 3, 9, 20, 29, 30 να τις καταψηφίσουμε και να κρατήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες A και B. Ευχαριστώ όλους τους μετέχοντες, ειδικά τους ε, σκιώδες για την ε, συνεισφορά τους. Αύριο θα ψηφίσουμε λοιπόν η Επιτροπή Ήτρε τον Οκτώβριο εκείνη. Και επιτέλους θα έχουμε και πάλι μια συζήτηση για τα κοινωνικά πολιτικά θέματα στην Ολομέλεια Σύνοδο του Νοεμβρίου. Θα το κάνουμε αυτό στο επίκεντρο και όχι στο περιθώριο. Εντάξει, χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό για το ότι τώρα έχουμε ένα άλλο κορυφαίο σημείο, τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη με τον Επίτροπο Άντορ. Βρίσκεται καθοδόν. Είναι στο διάδρομο ο κύριος Άντορ. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα λοιπόν. Θα τον περιμένουμε να έρθει, έτσι. Εντάξει, ωραία. Μέχρι να έρθει. Μάλιστα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Λάσλο Άντορ που είναι αρμόδιος για τα θέματα απασχόλησης, κοινωνικά θέματα και ένταξη και ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στο πλαίσιο του διαφρομένου διαλόγου, εμείς ε, ευρωβουλευτές μαζί του θα εξετάσουμε πολλά συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα. Έχουμε αρκετό χρόνο. Ναι, έτσι δεν είναι. Μέχρι τις 18.00 ε, ε, έχουμε χρόνο λοιπόν, περίπου μια ώρα. Προσβλέπουμε να ακούσουμε κύριε Επίτροπε. Το Ευρωκοινοβούλιο με ιδιαίτερη ευμένεια εισακούει και αφουγκράζεται αυτά που έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά ενδιαφερόμαστε για τις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Όπως συνηθίζουμε η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε την επόμενη περίοδο και θα μπορούσα να σκεφτώ λέγοντας ότι τώρα είμαστε στην τελευταία ε, χρονιά ε, που πριν από τις εκλογές, οπότε θα έπρεπε να μιλάμε λιγότερο και να ακούμε περισσότερο. Δεν θα πρέπει όμως να ηρωνευόμαστε γιατί η κρίση συνεχίζεται. Η ύφεση από ό,τι φαίνεται εδώ και μερικούς μήνες ήδη φάνηκε ότι κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη η ύφεση τελείωσε. Η δεύτερη ύφεση στην κρίση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια θετικά δείγματα ανάκαμψης Σημαίνει επίσης ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στην απασχόληση. Σε μερικές χώρες η ανεργία αρχίζει να μειώνεται. Κάτι που δεν περιμέναμε. Αυτά πάντως τα μικρά δείγματα βελτίωσης, τα δειλά δείγματα, δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε υπεραισιοδοξία. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Μπαρόσο, το αποσαφήνισε όταν ε, σας μίλησε για την κατάσταση πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πιστεύει ότι η κρίση θα τελειώσει γρήγορα. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας, ώστε να υπάρχει διώσιμη ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω απ' όλα, Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η στρατηγική ανάκαμψης περιλαμβάνει και σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής της νομισματικής ένωσης. Αυτό θα είναι και ένα από τα σημεία κλειδί που θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν μέσα στην επόμενη περίοδο. Θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Πάντως, θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι μια περίοδος κλειδί αυτή που διανύουμε τώρα και από την άποψη δημοσιονομικών αποφάσεων. Πόσο δηλαδή καθορίζουμε και σχεδιάζουμε τα δημοσιονομικά εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, και είναι σημαντικό για το δικό μου το χαρτοφυλάκιο, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συζητήσεις για τα δημοσιονομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για το Κοινωνικό Ταμείο και κάποια άλλα εργαλεία, συνεχίζονται οι συζητήσεις. Στο στάδιο αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική χρηματοδότηση της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής θα παραμείνει δεν θα διακινδυνεύσει και θα αποδώσει όσο γίνεται περισσότερο βάσει των προηγούμενων προτάσεων και διαπραγματεύσεων. Αυτό αφορά και το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Επιπτώσεων από την Παγκοσμιοποίηση, όπου οι παράμετροι δεν είναι τόσο ποσοτικοί όσο ποιοτικοί. Υπάρχουν και μερικά άλλα ζητήματα. Το πρόγραμμα αρρωγής προς τους ε, άπορους. Σήμερα επήγει το ζήτημα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν. Σε μερικές περιπτώσεις για τα προγράμματα απασχόλησης των νέων, που είναι μέρος της εγγύησης για τους νέους, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τελικοί διακανονισμοί καθυστερούν και τα πρακτικά βήματα προετοιμασίας. Ελπίζω όμως ότι εφ' εξής, πολύ γρήγορα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των χωρών μελών και των περιφερειών ελπίζω ότι θα επιταχυνθούν. Έρχομαι τώρα στο θέμα της νομισματικής ένωσης που είπα και πριν ότι είναι ένα στοιχείο κλειδί για τους επόμενους μήνες. Έχουμε ήδη συζητήσει μερικές φορές και ξέρετε ότι εκ παραλλήλου συζητάμε και στο Συμβούλιο με τους Υπουργούς και με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη. Το γεγονός ότι υπάρχει πόλωση. Φοβάμαι ότι από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας βλέπουμε ότι υπάρχει έντονα αυτή η πόλωση. Παρά την ανάκαμψη εξακολουθεί να υπάρχει πόλωση στον τομέα των κοινωνικών και της απασχόλησης. Γι' αυτό ετοιμάσαμε μία μεθοδολογία, νέα εργαλεία, τα οποία να μπορέσουν να βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά όργανα και το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να εντοπίζουν καλύτερα τις ανισότητες, τις ε, διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και να βοηθήσουν με προτάσεις για καλές λύσεις. Το θέμα της σύγκλησης τώρα. Η έννοια της σύγκλησης ίδια βρίσκεται στην καρδιά στον πυρήνα της κοινωνικής διάστασης των συνθήκων. Και άλλα όμως ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, όπως η στρατηγική για το 2020, πρέπει να ενισχυθούν. Συγχρόνως χρειάζεται μια εξισορρόπηση, δηλαδή να ενισχύουμε και την κοινωνική διάσταση για να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα μέσα στην κοινωνία, στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται έμφαση στην κοινωνική διάσταση μέσα στην Ευρωζώνη. Ο πρόεδρος Μπαρόσο έχει ήδη ανακοινώσει, έχει ήδη πει ότι τον Οκτώβριο θα γίνει αυτή η ανακοίνωση. Επιτρέψτε μου τώρα να σας δώσω ένα κατάλογο με κάποιους άλλους τομείς πάνω στους οποίους δουλεύουμε. Μήπως καταλήξουμε σε πρωτοβουλίες, οι οποίες είτε έχουν ήδη ανακοινωθεί, είτε πρόκειται να ανακοινωθούν εφόσον προηγουμένως κάνουμε τα βήματα που χρειάζεται και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει πριν τη λήξη της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομοθετικές προτάσεις. Προβλέπω την έγκριση κάποιων προτάσεων που βελτιώνουν τις προπτικές απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας, γιατί δεν έχει σημασία μόνο ο αριθμός των ε, θέσεων απασχόλησης, δεν είναι μόνο ο αριθμός που έχει πληγεί, αλλά και η ποιότητα της εργασίας και οι συνθήκες εργασίας δηλαδή. Είμαστε ουσιαστικά έτοιμοι με την πρόταση αυτή. Οδηγία για να επεκτείνουμε πέντε ε, οδηγίες που έχουν να κάνουν με τις θαλάσσιες μεταφορές. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση των υπηρεσιών απασχόλησης της Eurex διότι η κινητικότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αγοράς εργασίας, η ελευθερία ε, για να μπορεί κανείς να μπορεί να δουλέψει είναι μια βασική αρχή για μας. Πρέπει όμως να δούμε πώς θα στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία ακόμα περισσότερο για να μπορέσουν να υποφεληθούν αφενός οι άνεργοι και απ' την άλλη οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίε δεν βρίσκουν το κατάλληλο εργατικό δυναμικό στην περιοχή τους. Υπάρχει και μια άλλη πρόταση για ένα πλαίσιο ποιότητα όσον αφορά την ε, μαθητεία. Μετά από το προηγούμενο πακέτο που είχαμε τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Ένα άλλο πλαίσιο ποιότητα για την πρόβλεψη και την αναδιάρθρωση. Το δεύτερο θα βασιστεί στην ε, έκθεση που υιοθετήσατε εσείς ε, νωρίτερα μέσα στο 2013 για αυτό το θέμα. Υπάρχει μια πρόταση για μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ε, τη εργασία και την καταπολέμησή της. Η καταπολέμηση αδίλωτης εργασίας ε, ήταν αντικείμενο μιας διαβούλευσης που έγινε online και όταν ολοκληρώθηκε η διαβούλευση δεν έχουμε ακόμα, έχει ολοκληρωθεί μάλλον, αλλά δεν έχουμε ακόμα αποτιμήσει τα πορίσματα αυτής της διαβούλευσης. Κάποια από τα θέματα που σας ανέφερα, περιπίνει η αντίδοτη εργασία, η αναδιάρθρωση, η ενημέρωση και η διαβούλευση των εργαζομένων, ή ο κατακαιρματισμός αγοράς εργασίας, ε, τα θέματα του εργασιακού δικαίου και των συμβάσεων, θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο της διάσκεψης στα τέλη Οκτωβρίου για το εργατικό δίκαιο. Και φαντάζομαι θα τα ξέρετε όλα αυτά. Ξέρετε ότι σκοπεύουμε να διοργανώσουμε αυτή τη διάσκεψη τέλος Οκτωβρίου. Συνήθις ε, νομοθετική πρόταση είναι αυτή που συζητήθηκε πρόσφατα στο, στην Ορλομέλεια στο, το Σεπτέμβριο. Ήσασταν πολλοί από σας παρόντες. Το θέμα της ασφάλειας και της ε, υγείας στον χώρο εργασίας. Ε, και υπάρχει μια συνένεση για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής ε, γι' αυτό. Επίσης η επιτυχής δημόσια διαβούλευση μαζί με τις 500.000 συνεισφορές ε, προς το Σώμα των Επιτρόπων ε, είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Θα τα λάβουμε υπόψη μας για, το, για τα νέα βήματα. Για το 2014 τώρα. Κάτι που δεν θα είναι γεμάτη χρονιά ούτε για το Κοινοβούλιο αυτό, ούτε για την Κομισιόν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σταματήσουμε το έργο μας. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε προτάσεις που μπορεί να είναι σημαντικές. Η βασική νομοθετική πρόταση για το 2014 προβλέπεται ήδη στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν και είναι μια αναθεώρηση του κανονισμού για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλισης. Αυτή η πρόταση ίσως είναι ένα τμήμα ενό πακέτου κινητικότητας που θα προταθεί ε, στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν το 2014 και που θα αποτιμάει την κατάσταση και το πλαίσιο πολιτικής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Πέρα από αυτά, δεν σκοπεύω να προτείνω νέε νομοθετικέ πρωτοβουλίε που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν για το 2014. Όμω, πρότεινα να μπουν κάποιε ιδέε στο τραπέζι που έχουν το δυναμικό να δρομολογήσουν τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, να βελτιώσουν την κατάσταση απασχόληση και να συνεισφέρουν στην εμβάθυνση τη οικονομική και νομισματική Ένωση για την δημιουργία απασχόληση. Ε, οι μικροχρηματοδοτήσεις, ε, οι μικροπιστώσεις για τους επιχειρηματίες. Νομίζω ότι είναι έγκαιρη ε, πρωτοβουλία αυτή. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μια καλή ιδέα. Έχουν περάσει τρία χρόνια. Ας δούμε ποια ήταν η εμπειρία μαζί με όλα τα κράτη-μέλη και τα αντίστοιχα τα αρμόδια ιδρύματά τους. Ειδικά θέλω να δω τώρα με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση αυτή, αυτών των, αυτής της πρωτοβουλίας. Επίσης, ε, δημιουργεί θέση να απασχολεί στην πράσινη οικονομία. Αυτό εξετάζεται ε, σε την συγκρασία μεταξύ των υπηρεσιών μου και των υπηρεσιών της ε, Επιτρόπου Χέντεγκαρτ και του κ. Ποτότσνικ. Είναι χρήσιμο να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκίνησε το προσχέδιο για την... και ο δικός χάρτης για την εμβάθυνση της ε, Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και με μεγάλη χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Και θα ακούσω και τις επικρίσεις σας σε περίπτωση που έχετε. Ευχαριστούμε κρίσιμες αλλά και κριτικέ παρατηρήσει, αλλά και θετικού χαρακτήρα. Έχουμε ένα κατάλογο αγοριτών. Φτάσαμε ήδη στου 12. Κάναμε χρονομέτρηση για το χρόνο. Μετά από 6 που θα παρέμουν θα κάνουμε διάλειμμα. Θα απαντήσει ο επίτροπο και θα δούμε ποιο χρόνος απομένει. Δύο λεπτά όμω ανά κάθε ένα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε έτσι. Μπορούμε. Λοιπόν, α το κάνουμε. α ξεκινήσει το χρονόμετρο. Α, συγγνώμη, να σας πω ποιοι θα λάβουν τον λόγο. Ole Ludwigsson, das wären die drei, die sechs für die Αυτή είναι η πρώτη έξι. Haben wir Elisabeth Schröder, äh, Herr Plenkovic, Frau Maletic und der Thomas Mann. Das... είναι όλοι, οι δώδεκα. Α, συνεχίζεται ο κατάλογο. Ωραία. Θα παραμείνουμε στα δύο λεπτά. Α δοκιμάσουμε. Σάμπα Έρι, δύο λεπτά, όχι παραπάνω. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Αν θα, <clears throat> τον Οκτώβριο θα έχουμε την εκδήλωση να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Θα θέλαμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν έχουμε ακόμα μάθει τίποτα όσον αφορά τα όσα είπε ο κύριος Μπαρόζο. Ευελπιστούμε ότι στην ανακοίνωση που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπάρξουν κάποιες περισσότερες πληροφορίες που θα μας δοθούν. Ας εξετάσουμε τα διάφορα θέματα τα οποία αναφέρατε. Πίεζει πολύ ο χρόνος. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει πολύ χρόνο πια στη διάθεσή του. Εσείς λοιπόν αν θα εκπονήσετε μια πρόταση όσον αφορά την απασχόληση για εκείνους που εργάζονται ως ναυτικοί, θα πρέπει να τα καταφέρετε πολύ γρήγορα για να υπάρξει χρόνος να εξεταστεί η πρότασή σας. Έχουμε πολλές συζητήσεις που διεξάγονται για την χρηματοδότηση και να δούμε τι τελικά θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα χρηματοδώσει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα κάνει όσον αφορά τα κράτη-μέλη και τι θα χρηματοδοτήσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμή δεν αποσαφινίστηκε αυτό το θέμα, τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Θα είναι ευρωπαϊκά προγράμματα ή ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή θα είναι εθνικά προγράμματα τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν ακριβώ και θα δώσουν κίνητρα. Τι θα γίνει ακριβώ. Και τι θα γίνει όσον αφορά τα θέματα των συντάξεων. Δεν αναφέρατε τίποτα για αυτό το θέμα μέχρι στιγμή. Λοιπόν, Ποιε είναι οι απόψει σα για αυτά τα θέματα, Επίτροπε, ποιε είναι οι απόψει σα για τι ανάγκε αυτέ που υπάρχουν, οι λιγότερο ε, πλούσιοι, οι, εκείνοι που πιέζονται περισσότερο να μπορέσουν να έχουν κάποιες δυνατότητες. Είναι σημαντικό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε κάποιες πληροφορίε. Τι θα γίνει σε σχέση με την ε, αναδοχή εκδηλώσεων. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιο συμβιβασμό για εκείνους που θα αναλάβουν τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες. Έχετε κάποιο σενάριο. Τι θα γίνει σε σχέση με το hosting. Και επίσης όταν κάνουμε λόγο για στρατηγικές τι είναι εκείνο το οποίο προβλέπετε κύριε Επίτροπε. Θα μπορούσε να εξηγηθεί ότι υπάρχει ανάγκη να εκπονηθεί αυτή η στρατηγική όσο το δυνατόν ταχύτερα. Όλες οι πολιτικές ομάδες πιέζουν και θα ήθελαν να γνωρίζουν τι θα γίνει. Υπάρχει ανάγκη αυτή τη στρατηγική τώρα. Πρέπει να την εκπονήσετε και να την καταθέσετε το δυνατόν ταχύτερα. Αν πρέπει να πείσετε του συναδέλφου επιτρόπου σα, σα εύχομαι κάθε επιτυχία στο εγχείρημα. Θέλουμε η στρατηγική αυτή να κατατεθεί το δυνατόν ταχύτερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Σχεδόν τηρήσατε το χρόνο. Ο Αλεχάνδρο τώρα έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τόσα μας ανακοινώσατε και μερικά είναι καλά γιατί φαίνεται ότι θα προλάβουμε κάπως την καθυστέρηση που είχαμε μέχρι τώρα μετά από διάφορες υποσχέσεις που υπήρχαν. Τώρα υπάρχει και κάτι όμως το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο με την στρατηγική όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, δεν είναι ξεκάθαρο. Πότε ακριβώς το Σώμα των Επιτρόπων θα καταλήξει στη νέα στρατηγική. Και έχω και ένα σχόλιο για την κρίση, αναφερθήκατε στην κρίση. Πιστεύω κι εγώ ότι βλέπουμε στην άκρη του τούνελ λίγο φως. Αλλά το φως αυτό είναι το τέλος του τούνελ ή μήπως είναι κάποιο άλλο τα φώτα που βρίσκεται στην άλλη κατεύθυνση. Ο κόσμος δεν πάει καν να δηλωθεί και η απασχόληση λιγοστεύει. Ο κόσμος δεν πάει καν η κρίση. Δεν πρέπει να ερμηνευτεί από εσά, από τον Όλυ Ρεν, μακροοικονομικά. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε πόσοι δουλεύουν στην Ευρώπη σήμερα σε σχέση με αυτό που λένε οι στόχοι μας για το 2020. Για την ΟΝΕ τώρα. Ξέρω τις προσπάθειες που κάνετε και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε για να έχουμε δείκτες ώστε να ξέρουμε ποιες είναι οι διαφορές που υπάρχουν. Για να ξέρουμε και την πραγματικότητα. Όμως, δεν μας χρειάζεται μόνο να ξέρουμε ποιες είναι οι αποκλήσεις, θέλουμε να ξέρουμε και πώς θα τις διορθώσουμε. Η Ισπανία θέλει αυτόματους ε, σταθεροποιητές για να βγούμε από την κρίση, που να επικεντρώνεται στην απασχόληση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το αναλύει το φαινόμενο αυτό με μεγαλύτερη συνέπεια και προσφέρει εναλλακτικέ που δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί? Για πείτε μας και εσείς δύο λόγια γι' αυτό πριν φτάσετε στην ανακοίνωσή της Τέλος, για τη χρηματοδότηση. Μιλάμε για το κοινωνικό ταμείο, το ταμείο για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Μα εδώ διακυδεύεται η αξιοπιστία μας στους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να πετύχουμε λοιπόν και το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και οι πρωτοβουλίες για τους νέους μέχρι τα 30 να προχωρήσουν, γιατί έτσι θα έχουμε αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες, στους νέους κλπ. Κάτι το οποίο η Ευρώπη το χρειάζεται πάρα πολύ. Ευχαριστούμε λεπτά. Τώρα εσείς έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να έχετε δίκιο κύριε Επίτροπε ότι η συγκυρία θα συνεχιστεί με θετικό τρόπο μετά τις, από τις εκλογές στη Γερμανία. Κάτι άλλο ακούμε στη Γερμανία και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες και για τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν, δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης. Αλλά αν ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην Ευρώπη, έχουμε ατυπικές σχέσεις εργασίας, ε, παράνομη εργασία, κοινωνικό dumping, επισφαλή εργασία, περιορισμένου χρόνου εργασία, ελαστική εργασία, όλα αυτά δεν ελήφθησαν και δεν αντιμετωπίστηκαν με σοβαρότητα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια και καταλήξαμε σε αυτήν την κατάσταση. Σήμερα είδαμε και την κατάσταση ενός μιας τσεχικής εταιρείας, την Voxcom, όπου εργάζονται οι εργαζόμενοι εκεί για 120 ευρώ τον μήνα και από ξένες χώρες και από γειτονικέ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο θα έχουμε την έκθεση πρωτοβουλίας για τον έλεγχο εργασίας για αυτούς τους εργαζόμενους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νόμιμα εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις θα μπορούν να υποστηρίζονται και να υποστηρίζονται οι επιχειρήσεις. Θα έχουμε τους ελέγχους εργασίας και τους επιθεωρητές εργασίας που θα διαδραματίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει μια πλατφόρμα, μια πλατφόρμα κατά της παράνομης εργασίας τίθεται το ερώτημα για μένα. Πάει αρκετά μακριά αυτή η πρωτοβουλία. Δεν θα έπρεπε ευρωπαϊκή σε επιθεωρήσεις και ευρωπαϊκοί έλεγχοι να γίνονται. Στην αναζήτηση στοιχείων για την έκθεσή μου διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη είναι ανήμπορα να κάνουν κάτι λόγω του ότι δεν υπάρχει ανταλλαγή στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει εδώ ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και ευρωπαϊκά όργανα να δραστηριοποιηθούν με μεγαλύτερες εξουσίες. Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες μας στην Ευρώπη, τους εργαζόμενους γυναίκες και άντρε που έχουν εξοργιστεί πάρα πολύ για το κοινωνικό ντάμπινγκ, για το μισθολογικό ντάμπινγκ για τον ε, ε, ανταγωνισμό όσον αφορά για παράδειγμα ε, τα φορτηγά. Παίρνουν 300 ευρώ εκείνοι που εργάζονται σε αυτού του είδους μεταφορές. Δεν μπορούν να ζήσουν με αυτού του είδους μισθούς. Εδώ καλείται η Ευρώπη να δραστηριοποιηθεί και να βρει κανόνες και διατάξεις με, τις, με τους οποίους θα λειτουργεί αυτά. Ο Ούλε Κρίστενσεν έχει τον λόγο. Επόμενος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης, ε, λέει ο κύριος Κρίστανσεν και τον κύριο Επίτροπο για την έκθεση ε, πεπραμένων που μας έδωσε. Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Είναι σωστό και σημαντικό σε αυτόν τον τομέα να εκπονούμε, να εκπονήσουμε μια στρατηγική από πλευράς μας. Διότι κοστίζει πάρα πολλά χρήματα στα διάφορα κράτη-μέλη η αδράνεια και η απουσία ε, πρωτοβουλειών. Και έχουμε πολλά ατυχήματα στους χώρους εργασίας. Πολλοί αποβιώνουν κιόλας, πεθαίνουν άλλοι ασθενούν και θέλουμε εκείνοι οι οποίοι έχουν μια θέση απασχόλησης και θέλουν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας να μπορούν να το πράξουν. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την πτυχή της ασφάλειας και την προστασία των εργαζομένων περισσότερο. Φοβούμαι ότι η πορεία μπορεί να καταλήξει σε προς άλλη κατεύθυνση δυστυχώς. Και έχω και ένα παράδειγμα σε σχέση με τα όσα άκουσα για τους εργαζόμενους και εκπροσώπους από το επάγγελμα των κομωτών και κουρέων τι άκουσα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει σύντομα θα τοποθετηθεί σχετικά για τους κινδύνους αυτούς, για τη συμφωνία αυτή την οποία, ε, στην οποία συμφώνησαν οι κοινωνικοί εταίροι. Πρόκειται για πάρα πολύ επικίνδυνες χημικές ουσίες ε, στον τομέα του επαγγέλματος των κομμωτών ε, και θα ήθελα να γνωρίζω από εσά αληθεύουν αυτά. Αυτά τα στοιχεία είναι αληθινά και γιατί τώρα αυτή η μισθολογική συμφωνία, η σύμβαση αυτή θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο περαιτέρω. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Edith Μπάουερ, παρακαλώ Edith. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρει πολύ σύντομε ερωτήσει που σίγουρα μπορούν να ταιριάξουν και να ενταχθούν σε ένα λεπτό. Ε, η πολλοποίηση, η, η πόλωση είναι ε, έντονη και θα χρειαστούν νέα μέσα και νέα εργαλεία. Ποια μέσα και εργαλεία έχετε υπόψη να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ώστε να τερματιστεί η πόλωση η οποία όλο και οξύνεται στην Ευρώπη. Ερώτηση παριθμών 2 αφορά την εγγύηση για την νεολαία, για τους νέους. Τι είναι εκείνο το οποίο επιθυμείτε και προτίθεστε να κάνετε σχετικά με αυτή την εγγύηση για να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία αυτή να υποστηριχθούν τα άτομα, οι μαθητές οι οποίοι δεν συνεχίζουν τη σχολική τους εκπαίδευση και εγκαταλείπουν τη σχολική εκπαίδευση και μένουν στο περιθώριο. Τι θα γίνει, θα υπάρξει κάποια χρηματοδότηση, θα δοθούν κίνητρα, θα συνεχιστεί μέχρι το 30 έτος ε, υποστήριξη ώστε να μπορούν οι νέοι που είναι άνεργοι να υποστηρίζονται μέχρι το 30 τους έτος της ηλικία τους. Και τέλος, κοινωνικά συστήματα και κοινωνικά συστήματα ασφάλισης βέβαια που πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους και πρέπει να θεωρηθούν αυτά, να επανεξεταστούν από εσάς. Τι θα γίνει, θα αντικατασταθεί η 883 με κάποια νέα οδηγία και αν ναι, ποια μορφή θα πάρει αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Όλε Λούντβιξον, έχετε εσείς τον λόγο, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι ωραίο και καλό να έχουμε εδώ τον Επίτροπο ανάμεσά μας στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Σίγουρα. Αυτά τα οποία συζητούμε εδώ ανήκουν στα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες σήμερα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και από ίδια πείρα γνωρίζω ότι όταν η οικονομική συγκυρία θα βελτιωθεί παρόλα αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν άνθρωποι που θα βρίσκονται στις ουρές ε, ως άνεργοι και θα περιμένουν να βρουν μια θέση εργασίας και δυστυχώς θα κρατήσει περισσότερο αυτό το διάστημα παράδειγμα και δύο χρόνια. Είμαι πεισμένος ότι αν στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί μια καλή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και με τους οικονομικά εμπλεκόμενους στις αγορές εργασίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Γνωρίζω φυσικά ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που στοχεύουν, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ερώτημα, πότε όλα αυτά θα ξεκινήσουν και θα δρομολογηθούν ώστε να ολοκληρωθούν. Είμαστε πρόθυμοι να διεξαγάγουμε συζητήσεις με τους διαφορετικούς ε, κοινωνικού κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες για να εξευρεθούν λύσεις. Διότι δεν μπορούμε μόνοι μας να τα καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία με τους ε, ε, κοινωνικούς εταίρους, με τα συμβαλόμενα μέρη για συλλογικέ συμβάσει, εργοδότες και εργαζόμενους. Και τα συνδικάτα φυσικά εξίσου πρέπει και αυτά να εμπλέκονται και να συμμετέχουν στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και αυτό ισχύει για κάθε χώρα ξεχωριστά. Ο χρόνος, η χρονική στιγμή και συγκυρία έχει οριμάσει πλέον. Είμαστε στο 12 παρα 5. Πρέπει κάτι επιτέλους να κάνουμε, διότι όλα αυτά κράτησαν πολύ χρόνο και τώρα πρέπει να αναλυθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτά θέλω να μου πείτε επίτροπε. Τι προτίθεστε να κάνετε, τι έγινε μέχρι σήμερα και όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, που σήμερα αυτό είναι το μείζον, το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα τα άλλα προβλήματα. Παρότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό βέβαια. Ευχαριστώ. Είσαι κύριε, τελευταίο και μετά θα λάβετε εσείς κύριε Επίτροπε τον λόγο. Έχετε τον λόγο συνάδελφε. Ευχαριστώ. Ο Κροάτης συνάδελφος. Σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μου δώσατε τον λόγο και έτσι θα δραχθώ τη ευκαιρία, λέει ο κύριος Πλένκοβιτς, να παρέμβω. Υπάρχει η διερμηνία από τα κροατικά, έτσι, βέβαια υπάρχει. Πολύ καλά. Λοιπόν, Λοιπόν, Ω Ευρωβουλευτής ε, τη Επιτροπής ε, προπολογισμών με ενδιαφέρει πάρα πολύ το τμήμα των τοποθετήσεών σας όσον αφορά τα νομοθετικά μέτρα για το επόμενο δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο και την εγγύηση για τους νέους εξάλλου που είναι ένα τμήμα αυτών των δράσεων. Η Κροατία είναι ένα νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μια χώρα με πείρα όσον αφορά την ανεργία των νέων η αλήθεια είναι ότι οι νέοι μέχρι 24 έτη έχουν τεράστια προβλήματα να βρουν θέση εργασίας και έχουμε πάρα πολλούς ε, άνεργους, μακροχρόνια άνεργους. Χωρίς αμφιβολία θα θέλαμε εσείς πάντα να λαμβάνετε υπόψη το πρόβλημα της ανεργίας των νέων όταν στρέφεσαι στους πολίτες της Κροατίας ε, και ε, τοποθετήστε σχετικά. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα ένα τμήμα στην απάντηση αυτών των προβλημάτων είναι η εγγύηση για τους νέους. Μια συνέπεια του ότι η Κροατία είναι σήμερα ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, πριν από κάποια χρόνια και η χώρα σας είχε κάνει κάποια πειράματα και δοκίμασε λύσεις για εκείνους τους εργαζόμενους που εργαζόντουσαν στα σύνορα της Κροατίας για παράδειγμα. Τι βλέπουμε με αυτούς. Τώρα τα σύνορά μας με την Σλοβενία και με την Ουγγαρία ακριβώς δεν έχουν πλέον τελωνιακούς ελέγχους, δεν υπάρχουν τελωνιακοί. Εκείνοι που εργαζόντουσαν στα τελωνία είναι τώρα πλέον άνεργοι σε αυτά τα σημεία. Ήρθα σε επαφή μαζί μου επίσης ε, για να δουν πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνεργοι τελωνιακοί από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και φέτος και το επόμενο έτος 2014 τουλάχιστον να μπορέσει να δοθεί κάποια αποζημίωση, κάποια αντιστάθμιση ή να καταρτιστούν και να εκπαιδευτούν ώστε να βρουν νέα θέση απασχόλησης. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ξέρω συνάδελφε, είναι πολύ στενό το όριο, αλλά τα καταφέρατε, το τηρήσατε σχεδόν. Αγαπητέ Επίτροπε, έχετε τον λόγο, μπορείτε να λάβετε τον λόγο για μεγαλύτερο διάστημα, παρακαλώ. Ε, well, I hope I can... Θα προσπαθήσω να απαντήσω και δεν ξέρω τι άλλο έχετε να πείτε οι υπόλοιποι, γιατί τόσα πολλά είπαν ε, αυτή η πρώτη ομάδα ευρωβουλευτών για την ανεργία των νέων. Σχεδόν όλοι το θίξατε αυτό το θέμα. Τώρα φαίνεται λιγότερο ε, αυτό το πρόβλημα από ότι την Άνοιξη, γιατί τώρα έχουμε την εφαρμογή. Την Άνοιξη έχουμε τις συστάσεις του, της Συνόδου Κορυφής, ε, ε, είχαμε τη σύνοδο κορυφής που φιλοξένησε η Άγγελα Μέρκελ και συζητήθηκε πολύ σε αυτήν το, το θέμα. Ε, δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα. Τώρα πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή. Τον Οκτώβριο η Κομισιόν θα κάνει μια συνάντηση για τους ειδικού. Μέχρι τώρα όλα τα κράτη-μέλη είχαν έναν υπεύθυνο ε, υπάλληλο για την εγγύηση των νέων για το πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει σταματήσει. Για πολλές χώρες, όπως και την Ιταλία και την Πορτογαλία, η Κομισιόν βοηθάει τις αρχές για να ετοιμάσουν το εθνικό σχέδιο για την εγγύηση των νέων. Και ο αρμόδιος επίτροπος θα πάει για να συζητήσει διμερώς με, τους, με τις αρχές των χωρών αυτών το σχέδιο. Στη συνάντηση λοιπόν του Οκτωβρίου η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης θα διευκρινίσει με κάθε χώρα που βρίσκεται τι έχει, τι έχει ε, σχεδιάσει κάθε χώρα, γιατί οι 20 χώρες που ε, εποφελούνται από αυτήν την πρωτοβουλία για την εγγύηση των ε, νέων θα πρέπει να είναι έτοιμες και να έχουν τα σχέδιά τους ολοκληρωμένα μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Οι υπόλοιπε αργότερα. Από πού προέρχονται τα λεφτά. Τα λεφτά Ε, προέρχονται από τρεις διαφορετικούς πόρους. Εθνικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τους ε, νέους σε συγκεκριμένες όμως περιοχές. Το τελευταίο θέμα είναι ευαίσθητο, γιατί η ομάδα στόχος και, ομα... και οι περιοχές στόχος δεν έχουν αποφασιστεί. Συζητηθούνται ακόμα και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Εγώ μπορώ να σας εξηγήσω τη δική μας αρχική πρόταση. Δεν έχουμε αιμονή με το νούμερο 25, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι αν ε, έχουμε ένα νέο εργαλείο που θα είναι διαφορετικό, θα κάνει τη διαφορά, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις χειρότερες, στις πιο πληγήσεις περιοχές. Γι' αυτό είπαμε μέχρι 25. Αν όμως κάποιος έχει καλύτερη ιδέα, το συζητήσουμε. 20 θα ήταν γελίο, γιατί τότε το όλο εργαλείο αποδυναμώνεται και αυτοί που το χρειάζονται, αυτοί που χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια, δεν θα την πάρουν. Για το θέμα του ορίου ηλικίας. Γιατί είπαμε μέχρι 25 χρονών. Γιατί η λογική της εγγύησης ε, για τους νέους είναι να βοηθήσει τη μετάβαση των νέων από το σχολείο στην ε, απασχόληση. Αυτοί που σταματάνε το σχολείο νωρίς να μπορούν να βρίσκουν μια πρώτη θέση. Θα έχουν λοιπόν μια εξατομικευμένη ε, βοήθεια, ειδικά αν προέρχονται από μειονεκτούσες ε, οικογένειες και περιοχές. Είναι δύσκολο να βρει κανείς... Ε, είναι δύσκολο να βρει κανείς δουλειά λοιπόν αμέσως όταν αντιμετωπίζει πολλές δυσχέρειες. Γι' αυτό αρχικά εστιαστήκαμε λοιπόν από πλευράς Κομισιόν στο όριο των 25 ετών. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας και πόσους πόρους έχουμε για να χρηματοδοτήσουμε αυτό το σχήμα. Αν είχαμε περισσότερους πόρους θα μπορούσαμε να είχαμε επεκτείνει αυτό το εργαλείο σε πιο, μεγάλα, πιο ηλικιωμένα άτομα. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε στα 30 ας πούμε. Φυσικά λόγω της δύσκολης κατάστασης με την απασχόληση ορισμένες χώρες θα ήταν δικαιολογημένο αλλά υπάρχουν και διαφορές ε, ως προς τη διάρκεια του σχολείου. Σε ορισμένες χώρες ε, ο κόσμος βγαίνει από το εκπαιδευτικό σύστημα αργότερα από ό,τι σε άλλες. Ορισμένες επίσης χώρες έχουν και την τάση ε, αμέσως με το σχολείο να στέλνουν τον κόσμο στο χώρο απασχόλησης και μετά να ξαναπηγαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ άλλοι αμέσως με τη δευτεροβάθμια πάνε στην τριτοβάθμια. Υπάρχουν διαφορές λοιπόν. Αν όμω θέλαμε να καλύψουμε περισσότερο, θα πρέπει να είχαμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Στην ε, επερχόμενη επίσκεψή μου στην Κροατία, κύριε Πλάνκοβιτς, θα συζητήσω με διάφορους υπουργούς, διάφορους αρκετούς υπουργούς, το θέμα της, ανα... της απασχόλησης των νέων. Όταν εντάχθηκε η Κροατία, ήταν η τρίτη χώρα ως προς την ανεργία της. Θα συζητήσω με διάφορους υπουργούς την ανεργία των νέων. Θα συζητήσω επίσης και το σχήμα αυτό, αλλά και το θέμα χρηματοδότησης. Άκουσα τόσες ερωτήσεις και για την νομοθεσία πολλές και ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες να υπάρξει μια σύγκληση για την απόσπαση των εργαζομένων. Η Ιρλανδική Προεδρία έκανε, Προεδρία έκανε ό,τι μπορούσε και η Λιθουανική επίση κάνει ό,τι μπορεί, ούτω ώστε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βρουν κοινή θέση. Και εγώ ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη προσωπικά να καταλάβουν τα επιχειρήματα των άλλων κρατών μελών. Ορισμένα κράτη-μέλη έδειξαν μια κάποια ευελιξία. Πρέπει να το πω αυτό ενώ κάποια άλλα όχι. Ο συμβασμός είναι εφικτός μόνο όταν ε, κάνει ο καθένας μια χειρονομία και καταλάβει λίγο τον άλλον. Και υπάρχει μια σύγκληση λοιπόν έτσι. Ελπίζω να καταστεί εφικτό αυτό. υπάρχουν περιπτώσει όπου δεν έχουμε νέα νομοθεσία και υπάρχουν πολλές προσφυγέ στα δικαστήρια. Ε, τα δικαστήρια αποφασίζουν τελικά για την, τα θέματα απόσπαση εργαζομένων και ειδικά αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν πάρα πολύ την απόσπαση νέων εργαζομένων για την μεταφορά συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Ο τριμερή διάλογο ξεκινάει σήμερα. Ρώτησα κάποιο βουλευτές πότε ξεκινάει σήμερα. Και ελπίζω ότι, ότι αυτός ο πολύ σημαντικός φάκελος θα διεκπεριωθεί γρήγορα. Κυρία Μπάουερ, ρωτήσατε για το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας μας για του χρόνου. Ετοιμάζουμε μια αναθεώρηση για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα έγγραφο της κυρίας Ρέντινγκ που δημοσιεύτηκε το Μάιο. Ε, Ετίθενταν διάφορα ερωτήματα εκεί. Πόσο καιρό ε, ένα άτομο μπορεί να παίρνει επίδομα ανεργίας από τη χώρα προέλευσή του να αλλάζει χώρα. Σήμερα, α πούμε, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 3 με 6, 3 ε, με 6 μήνε. Όταν έχουμε μεγαλύτερη κινητικότητα στο μέλλον, έχει νόημα να παρατείνουμε αυτή την περίοδο, να μεγαλώσει αυτή η περίοδο, ή να θέσουμε ένα νέο πρότυπο στην Ευρώπη. Τέτοιου τύπου ερωτήσει ε, μπορούν να απαντηθούν με το διάλογο. Άκουσε αυτά που είπε ο κύριος Ερή. Για την πρόταση που πρέπει να κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν θα προσπαθήσουμε κύριε Ερή. Μπορώ να συνεχίσω. Η κοινωνική διάσταση, εντάξει, πράγματι η πόλωση είναι μείζον ζήτημα εδώ. Και το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια συστημική ικανότητα να εποπτεύσουμε αυτή την πόλωση με ένα ε, σύνολο δικτών ε, που θα μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την πόλωση, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα διαδραματίζουν ένα πιο ενδυναμωμένο ρόλο. Ο κύριος Σέρκας ε, στο ίδιο πλαίσιο μίλησε για τους αυτόματους σταθεροποιητές. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ότι διεξήγαγε ήδη συζήτηση για την εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων το Ευρωκοινοβούλιο. Θα συμμετάσχω με το Ίδρυμα Bertelsmann, Bertelsmann Foundation σε μια τέτοια εκδήλωση για τις εναλλακτικές δυνατότητες για τέτοιου είδους δείκτες. Γνωρίζω το IMF, το έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ένα τέτοιο μέσο αναφέρεται στο σχέδιο αυτό, στο blueprint. Είναι λοιπόν συνάδει και είναι συμβατό με την ε, πορεία που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι όμως πρόεινο να πούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα δύο λεπτά θα τα καταφέρουμε τώρα με τους επόμενους. Η κυρία Ελίζα Μπεσρόιντα, δύο λεπτά. Μάλιστα. Προσφέρεται λοιπόν εδώ αυτό το οποίο είπατε. Να συνεχίσω κύριε Επίτροπε ε, Άντορ με την κοινωνική διάσταση. Έχουμε την νομισματική ένωση, έτσι. Κατάλαβα καλά αυτό που προπαρασκευάζεται φέτος ακόμα θα είναι το stabilizator, δηλαδή δεν σας συμπεριλαμβάνεται αυτό, δεν θα υποβάλλετε πρόταση για τους σταθεροποιητές, ε, για τη σταθεροποίηση. Είναι εκείνο το μέσο το οποίο θα επέλυε το ζήτημα που είναι θέμα κλειδί. Δηλαδή αν θα έχουμε κοινωνική και οικονομική και οικολογική ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των, της ε, νομισματικής ένωσης και των πυλώνων της και των στοιχείων της. Έχουμε μια μη ισορροπή σχέση και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να τοποθετηθείτε εξειδικευμένα. Θα υπάρξει πρόταση για σταθεροποιητή στην πρόταση που θα υποβάλλετε και πότε θα, κατα, θα κατατεθεί και θα δημοσιοποιηθεί. Επίσης για το θέμα πότε θα δημοσιευθεί με ενδιαφέρει πρόταση που κάνατε για μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της παράνομης ε, εργασίας. Τι ακριβώς θα υποβάλλεται ως πρόταση και ποια μορφή και διατύπωση θα έχει και πότε θα ε, υποβληθεί η πρότασή σας. Με ενδιαφέρει επίσης και όσον αφορά και ένα πράγμα όπου αναμένουμε μεγάλο χρονικό διάστημα γι' αυτό. Είναι το ποιοτικό πλαίσιο για τους ασκούμενους. Είπατε το Δεκέμβριο θα υποβάλλετε κάποια πρόταση. Ποια πρόταση θα είναι αυτή. Θα είναι πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου. Θα γίνει όπως ε, έγιναν προηγούμενα τα πράγματα με την εγγύηση για τους νέους, για την νεολαία ή ποια άλλη μορφή θα πάρει. Ένα τελευταίο σημείο θέλω να αναφέρω για το οποίο χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι η πρωτοβουλία σας για clean jobs, καθαρές θέσεις εργασίας και απασχόλησης. Ποιο μήνα θα υποβληθεί. Τώρα σύντομα θα την υποβάλλετε. Διότι είναι μια πρωτοβουλία που απέρευσε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επιθυμούμε ουσιαστικά μέσα σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία που θα είμαστε αρμόδιοι ως Ευρωβουλή να υποβληθεί από εσά ώστε να μπορέσουμε να ε, οδηγήσουμε αυτή την πρόταση σε αίσιο πέρα. Σας ευχαριστώ. Η Ντανούτα έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρε ευχαριστώ. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τα δύο λεπτά είναι πάρα πολλά για μένα. Επίτροπε, Ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε σήμερα. Όμως πολύ λίγα μας είπατε για το τι προτίθεται και τι σχεδιάζει να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τους επόμενους μήνες. Εγώ και οι συνάδελφοί μου θα θέλαμε σήμερα ήδη να γνωρίζαμε τι θα συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι θα αναγνώσουμε σε αυτήν για την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Θα ήθελα να ακούσω κάτι παραπάνω για αυτά τα θέματα. Η ερώτησή μου τώρα. Πώς επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει τις δαπάνες όσον αφορά το κοινωνικό ταμείο και πώς θα υποπτεύει αυτές τις δαπάνες ουσιαστικά από πλευράς της. Και τέλος, πώς ε, θα διαμορφωθούν τα προγράμματα και θα λειτουργήσουν τα προγράμματα για την υπέρβαση της κρίσης, την αντιμετώπιση της κρίσης και τι θα γίνει με την ε, εγγύηση των νέων, για τους νέους. Πώς θα υποπτευθούν όλα αυτά. Η μέχρι σήμερα πείρα μας ήταν μάλλον αρνητική. Οι εμπειρίες μας ήταν αρνητικές. Τα διαθέσιμα κονδύλια δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε. Σύντομα θα έχουμε περισσότερα κονδύλια στη διάθεσή μας. Οι ευθύνε μας θα είναι έτσι μεγαλύτερες λοιπόν. Η επόμενη ερώτησή μου αφορά την απόσπαση εργαζομένων για τους αποσπόμενους εργαζόμενους. Πώς έχουν τα πράγματα, τι σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα διότι πρέπει πραγματικά να εξευρεθεί ένα συμβιβασμός από το Συμβούλιο. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συνεισφέρει από πλευρά του, ώστε να εξευρεθεί ένας τέτοιος συμβιβασμός που θα είναι συνετός. Η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια που δημιουργείται για τους ε, ευρωβουλευτέ σε σχέση με τα θέματα της απόσπασης ε, για τους εργαζόμενους είναι μεγάλο πρόβλημα. Να προσθέσω κάτι. Στην Πολωνία ένα πιλωτικό σχέδιο υλοποιείται. Μία ειδική δημογραφική ζώνη. Σε κάποιες περιφέρειες κάποιες δραστηριότητες ε, ασκούνται και υλοποιούνται για να ξεπεράσουμε προβλήματα, να υπερβούμε τα προβλήματα και της Πολωνίας και της Ευρώπης. Για τα δημογραφικά προβλήματα που θέλουμε να αντιμετωπιστούν. Τον Μάρτιο προβλέπεται μια σύνοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε να παρουσιαστείτε και εσείς και να συμμετάσχετε σε αυτήν. Ευχαριστώ. Πολλές συνόδους θα έχετε επίτροπε και συμμετέχετε σε αυτές. Ε, εσείς παρακαλώ δύο λεπτά. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, hvala lijepo e, povjereniku na... Što? E, ono što bi ja για την παρουσίασή σας και για την, uh, τις απαντήσεις σας. Θέλω να αναφερθώ στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Υπάρχει εδώ πέρα μια σημαντική πρόκληση και είναι ο συνδυασμός διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων για ένα και το ίδιο μέτρο για ένα και τον ίδιο σκοπό. Μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα το νέο αυτό δημοσιονομικό μοντέλο. Το γεγονός δηλαδή ότι σε περιπτώσεις κρίσης προσπαθούμε να καινοτομήσουμε και να δούμε πώς θα συνδυάσουμε μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της εκπαίδευσης. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έγινε κατάφορη αυτή η ανάγκη του συνδυασμού των κονδυλίων. Ελπίζω ότι ο Επίτροπος Αντόρ μαζί με τον Επίτροπο Χαν θα μπορέσουν να βρουν νέους τρόπους για να συγκεντρώσουν όσο γίνεται περισσότερα κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αντλήσουν και επιπλέον κονδύλια από το κοινωνικό ταμείο για την κατάρτιση, κάτι που είναι τόσο αναγκαίο προκειμένου να μπορέσουν να βρουν ε, δουλειά οι άνθρωποι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δημιουργηθούν μέσω του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει κάνει με την ειδίκευση μέχρι το 2020, την ευφύ που απαιτεί νέες μονάδες, οι μικρές, ε, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις όμως που ασχολούνται με αυτά και άλλοι φορείς πρέπει να παρουσιάσουν κάποια τεκμηρίωση. Εσείς πώς βλέπετε να τίθεται στην πράξη αυτή η εταιρική σχέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κοστέλο. Δύο λεπτά κι εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Κύριε Επίτροπε ένα σχόλιο και τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτον, είπατε ότι φτάνουμε στο τέλος της ύφεσης, αρχίζει η ανάκαμψη και στην Ελλάδα λέμε το ίδιο, όμως οι Τρόικα εξακολουθούν να δουλεύουν βάσει της λιτότητας, είναι τζάνκες της λιτότητας. Η δημοσιονομική στόχη όμως, τι είναι, 3,1 δισεκατομμύρια να βγουν από την οικονομία μας, ενώ θα μπορούσαμε να το πετύχουμε με 2,5. 440 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από τον προπολογισμό μας για τα κοινωνικά εάν τηρηθούν αυτά που ζητάει η Τρόικα. Οπότε για την Ιρλανδία μπορείτε να το κάνετε στον επόμενο προπολογισμό. Έπειτα για την εγγύηση των νέων πρέπει να επιταχυνθεί το πρόγραμμα αυτό. Μιλάμε για προκαταβολές και όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει προτεραιότητα για τα χρήματα που θα είναι διαθέσιμα το 2014 και 2015. Μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τις προκαταβολές για την εγγύηση για τους νέους, αυτό το front loading για το 2014 και 2015 και ότι μπορούμε έτσι να προσφέρουμε στου ανθρώπους που τώρα είναι 23 να έχουν την ευκαιρία να υποφεληθούν πριν γίνουν 25 ή θα πάρει περισσότερο χρόνο. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν υπερβολμένο ακόμα περισσότερο. Επίσης, Επίτροπε, αναφερθήκατε στο πολιτικό πλαίσιο για τους ε, ε, ανθρώπους που βρίσκονται σε μαθητεία. Πρέπει να συνάδει αυτό να πηγαίνει χέρι-χέρι με την εγγύηση για τους νέους. Πότε θα έχουμε προτάσεις λοιπόν και πότε θα γίνει ο συγχρονισμός με την εγγύηση για τους νέους. Τέλος, είμαι συγγήτρια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτάσεις τις σχετικές με τα προγράμματα για τους νέους. Κύριε Επίτροπε, θα μπορέσετε να διασφαλίσετε στον κόσμο να τους εγγυθείτε ότι θα τους βρείτε ε, κάποια διέξοδο στο θέμα της απασχόλησης. Δύο λεπτά, Πατατσίνο. Ευχαριστώ. Κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό υποφελούμε από αυτή την ευκαιρία στην Επιτροπή αυτή, τώρα που είσαστε εσείς εδώ, για να σας ρωτήσω απευθείας κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την προσωρινή εργασία. κάτι το οποίο πλήττει τον ίδιο τον ιστό των οικογενειών και της κοινωνίας. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι υποφέρουν από κακές συνθήκες εργασίας, από συμβάσεις πολύ μικρού χρόνου, λίγου χρόνου, και έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους και να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Ρωτάω λοιπόν ποιος είναι ο επίσημος ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτής της λεγόμενης precarious work, της κακής ποιότητας εργασίας, προσωρινής εργασίας. Πώς θα αντιμετωπίσετε από την Επιτροπή αυτό το νέο φαινόμενο. Τι θα κάνει η Επιτροπή στην περίπτωση που κράτη-μέλη δεν καταπολεμούν το φαινόμενο αυτό. Και το λέω γιατί εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν κάτω από τόσο κακές συνθήκες είναι τελικά η φτωχή των κοινωνιών μας. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την Επιτροπή να μου πει τι σχέδια έχει. Πώς θα βοηθήσουμε 20 εκατομμύρια ανθρώπους να βγουν από την ένδια μέχρι τα τέλη του 2020. Τέλος, μπορείτε να μας δώσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. για την οδηγία όσον ε, αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται στις θαλάσσιες μεταφορές. Πότε θα είναι έτοιμη αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Η δική μου παρέμβαση και οι δικές μου ερωτήσεις ε, από τα όσα επεξηγήσατε ήδη καλύφθηκαν εν μέρη σε σχέση με την χρήση των πόρων στις, πιο, ε, στις ιδιαίτερα πλη, πληττόμενες περιοχές από την ανεργία των νέων και θα ήθελα αυτό ε, να αναφέρω ότι χαιρετίζω αυτή την, αυτό το σθένος ε, και αυτό τον ορισμό μέχρι το 24ο έτος να βοηθήσετε τους νέους και την ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευτικά όσον αφορά τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη για την πρωτοβουλία για τους νέους όπως στην περίπτωση της Πορτογαλίας π.χ. Τούτων λεκτέντων όμως θα ήθελα από πλευράς μου να ζητήσω από τον κύριο Επίτροπο κάτι στο πακέτο μέτρων για την κινητικότητα την εργασιακή που σκοπεύετε να παρουσιάσετε το επόμενο έτος να λάβετε υπόψη ένα σημαντικό φαινόμενο το οποίο επίσης συμβαίνει στις νότιες χώρες της Ευρώπης που επίσης συναρτάται με την ανεργία των νέων και είναι ότι υπάρχουν νέοι με προσόντα, από τους πιο προσοντούχους όλης της Ευρώπης που φεύγουν από τις χώρες μας. Η διαρροή των νέων, brain drain, διαρροή εγκεφάλων, ε, φεύγουν, μεταναστεύουν και αναζητούν απασχόληση αλλού. Αυτό είναι εις βάρος της Ευρώπης. Εδώ θα μπορούσε ίσως να εντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα θετικό πλαίσιο για να ευνοηθεί η επιστροφή αυτών των νέων στις χώρες τους. Το άλλο θέμα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα προβλήματα στην ε, απάντηση στην ε, ανεργία συνολικά και στην ανεργία των νέων ειδικότερα. Τι είναι εκείνο το οποίο θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνενώσει τις προσπάθειες στο συλλογικό σώμα των επιτρόπων για να ευνοήσει την χρηματοδότηση αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ευνοηθεί η δράση υπέρ των νέων. Ευχαριστώ. ο Μαν. Α, αποσύρει την παρέμβαση. Μία ερώτηση τώρα. Κύριε Επίτροπε, η εμπειρία σας με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ποια είναι έχει εγκριθεί από τα κράτη-μέλη. Συμφωνείται από τα Ευρωπαϊκά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι παραπάνω από τον ένα συντονιστή, να κάνει κάτι παραπάνω, να συλλέξει δεδομένα και να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να δραστηριοποιηθούν με βάση αυτά τα στοιχεία. Χρειάζεται κάποιο χρόνο. Ήταν η τελευταία μα ερώτηση. Περνάμε τώρα στο ρολόι. 15 λεπτά έχετε αγαπητέ Επίτροπε, με πάρα πολλέ, απίστευτα πολλέ ερωτήσει. Προσβλέπουμε να δούμε στα 15 λεπτά πώ θα απαντήσετε και θα καλύψετε. Ολοκληρώνουμε και αύριο μετά θα έχουμε στις 9 η ώρα τη συνέχεια της συνεδρίασής μας γιατί θα κλείσουμε μετά τον Επίτροπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ερωτήματα τα οποία απέμειναν και από τον πρώτο γύρο και θα προσπαθήσω να επανέλθω και σε αυτά και πραγματικά να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν ε, όλα αυτά για να δοθούν απαντήσεις. Ίσως θα ήταν δύσκολο να απαντηθούν εξειδικευμένα όλα αυτά Καμιά φορά όταν έχουμε μια πρωτοβουλία που βρίσκεται απότερα χρονικά, αλλά καμιά φορά συμβαίνει και το αντίθετο. Αν είναι την επόμενη εβδομάδα να γίνει κάτι, θα πρέπει να ζητήσω να δείξετε την υπομονή σας και την κατανόησή σας να έχουμε, να εξεύρουμε αυτά τα στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία μας. Όμως πραγματικά τώρα στη συνέχεια, για παράδειγμα, από πλευράς να ε, ρωτήθηκε τι γίνεται με την κοινωνική διάσταση όσον αφορά την ανακοίνωσή μας και τι θα συμπεριλάμβανε η ανακοίνωσή μας ακριβώς. Ας αναφερθώ στην πρόσφατη εμπειρία μου στην ε, Πολωνία. Πήγα στο Κλίνιτσε για το οικονομικό φόρουμ και μετά είχαμε ε, εκδηλώσεις εκεί και για να σας δώσω μια σύντομη απάντηση. Συμφωνώ πάρα πολύ με την προσέγγιση του κυρίου Μπιελέτσκι, πρώην Πρωθυπουργού της Πολωνίας, με τον οποίο συναντήθηκα για αυτό το θέμα, ο οποίος ουσιαστικά τι είπε. Είπε αν η υποτίμηση είναι ο κύριος μηχανισμός προσαρμογής για την Πολωνία, τότε η Πολωνία θα πρέπει να προβληματιστεί πολύ περισσότερο γιατί αν θα, αν θα προσχωρούσε στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση ή όχι. Διότι όλες οι επιπτώσεις ε, σε σχέση με τη ζήτηση και τις επιπτώσεις μιας εσωτερικής υποτίμησης, όλες οι επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές. Και αυτό ήταν ένα από τα αναλυτικά επιχειρήματα πίσω από τη θέση αυτή την τοποθέτηση για την προβλεπόμενη πρόταση που εμπνέει αυτές τις αναλύσεις αλλά και την, τις απαντήσεις στο πολιτικό επίπεδο. Δεν θα υπάρξει βιασύνη, δεν θα προσπεράσουμε τις εξελίξεις αλλά για, σε σχέση με συγκεκριμένα νέα στοιχεία για την νομισματική ένωση πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο, ένα ευρύτερο εγχείρημα. Υπάρχουν και άλλα πολλά στοιχεία βέβαια τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν και να επιταχυνθούν για παράδειγμα αν θέλουμε να υλοποιηθούν όλα με ένα ταχύτερο τρόπο σε σχέση με τα όσα συνέβησαν κατά το πρώτο ήμιση του έτους. Όμως η κοινωνική διάσταση, η ανακοίνωση για την Δεν ήμουν σε θέση να σας δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία για την πρωτοβουλία όσον αφορά τους ναυτικούς. Και τα, στα λίγα λεπτά που πέρασαν δεν ε, βελτιώθηκαν τα πράγματα για να μπορέσω να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Δείξτε κατανόηση παρακαλώ λοιπόν. Κάποιες από αυτές τις αποφάσεις δεν έχουν ακόμα ληφθεί και δεν είναι έτοιμες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως από την άλλη πλευρά <clears throat> ουσιαστικά βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένη φάση των διαβουλεύσεων για την προπαρασκευή αυτής της ανακοίνωσης για τους ναυτικούς. Τώρα, αν η πλατφόρμα μας για την καταπολέμηση της παράνομης εργασίας θα επαρκεί και θα κατατεθεί έγκαιρα και είχαμε και άλλες ερωτήσεις συναφείς. Φυσικά <clears throat> όλα αυτά όταν θα έχουν οριμάσει θα γίνουν προσπαθούμε να δώσουμε feed-in, να εντάξουμε σε αυτή την πρωτοβουλία όλα τα στοιχεία τα οποία πορεύουν από τη διαβούλευση. Αυτός ήταν και ο σκοπός της διαβούλευσης εξάλλου. Να έχουμε ιδέες πρακτικής μορφής και πρακτικές ιδέες να προαχθεί και να εντείνουμε τη συνεργασία όσον αφορά τους ε, εργασιακούς ελέγχους, επιθεωρήσεις ε, όσον αφορά θέματα εργασίας ε, Τώρα για την προσδοκία αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν ε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ίδρυε επιθεωρήσεις εργασίας, όχι. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σκοπεύουμε να κάνουμε. Θέλουμε να υπάρξει μια καλύτερη βελτιωμένη ανταλλαγή στοιχείων και συνεργασίας και ενημέρωση σε σχέση με τους ε, ελεγκτές και επιθεωρητές εργασίας σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ο στόχος μας. Στην επίσκεψή μας στην ε, Ολλανδία και σε σχέση με τον Πρωθυπουργό, με εκείνον, εκείνον που είναι ε, με πρωτοβουλία του δημιουργήθηκε ο Orange Code όχι μόνο για τα θέματα μετανάστευσης, να μην υπάρξει παρανόηση, αλλά για τους όρους εργασίας και απασχόλησης των μεταναστών από μια τρίτη χώρα. Και αυτό είναι ουσιαστικό ζήτημα και πρέπει να τύχει της προσοχής μας. Εδώ υπάρχουν πολλέ δυνατότητε να διασφαλίσουμε καλύτερε συνθήκε απασχόληση, να τυποποιήσουμε και να επισημοποιήσουμε τι πτυχέ, τι συνιστώσει τη απασχόληση, καθώ επίση και τη διασφάλιση φορολογικών εσόδων όσον αφορά την απασχόληση τέτοιων εργαζομένων από τα κράτη-μέλη με εισφορέ κτλ. Είναι σημαντική στόχη αυτή που συνδέονται με αυτή τη μελλοντική πρωτοβουλία που θα αναλάβουμε. Τώρα από την άλλη πλευρά πράγματι είμαστε υπέρ τη κινητικότητα και την προάγουμε η ελευθερία να εργάζεται κάποιος σε μια άλλη χώρα πρέπει να είναι πάντα σεβαστός, σεβαστή δικαίωμα. Όμως βλέπουμε επίσης ε, τι είναι αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς ε, Ευρωβουλευτά. Η πιθανή ζημία που μπορεί να προκληθεί ίσως ε, σε κάποιες τρίτες χώρες. Αν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα <clears throat> έχουμε μεγάλη διαρροή δυναμικού από μια χώρα. Για παράδειγμα, έθιξα αυτό το θέμα όταν πήγα στη Λετωνία πρόσφατα που είναι μια χώρα <clears throat> που επενέθηκε για τις οικονομικές επιτυχίες της και την δυνατότητά της να ενταχθεί στο ευρώ ε, το 2014. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ε, δημοσιονομική εξυγίαση σε αυτή τη χώρα έγινε σε μια χρονική συγκυρία όπου πάρα πολλοί πολλοί νέοι αποχώρησαν και αν δεν ε, μπορούσε να αντιστραφεί αυτό θα ήταν μια μακροπρόθεσμη απώλεια σε σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο εις βάρος της οικονομίας διότι θα άλλαζε το ποσοστό εξάρτησης ε, και αυτό είναι μεγάλο σημαντικό στοιχείο για την κοινωνική ασφάλιση αν υπερβολική Κάπολοι από τους εργαζόμενους εγκαταλείψουν μια χώρα και πάψουν πια να συνεισφέρουν όσον αφορά και τα ταμεία και την ασφάλιση, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να υπάρξει ίσως ένα άνοιγμα ή ένα, ή ένα πλήγμα, μια, ένας κλειδονισμός. Πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά, πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει όχι μόνο μονόδρομος μετανάστευσης και αποχώρηση από αυτή τη χώρα, αλλά και επιστροφή κυκλικά, με, όπως και στην Ισπανία. Μετά από κάποια χρόνια, δύο-τρία χρόνια για παράδειγμα, μπορεί να σημειωθεί μια αντίστροφη φορά και να επιστρέψουν ε, πολλοί στην Ισπανία. Με τη δημιουργία της εγγύησης των νέων πρέπει να διασφαλίσουμε τη δημιουργία διάνοιξης ευκαιριών για αυτούς τους νέους στις χώρες τους. Γι' αυτό είναι τεράστια σημασία να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρωτοβουλία για την εγγύηση των νέων. Θα διασφαλιστεί ότι η πορεία εκτός μιας χώρας δεν είναι η μόνη δυνατότητα για όσους έχουν χάσει τις ελπίδες τους στη χώρα τους. Μπορούν να βασιστούν και στις τοπικές υπηρεσίες που θα είναι δικτυωμένες με τους κοινωνικούς εταίρους θα παρέχουν καλύτερες πληροφορίες ε, για τις διαθέσιμες ε, θέσεις απασχόλησης ή τις μελλοντικά διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης θα μπορούν να κινητοποιήσουν ε, την πρόσφατα στη διάθεσή τους οικονομική υποστήριξη ώστε να επιδοτούνται είτε θέσεις απασχόλησης είτε να επιδοτείται η κατάρτιση ή η μαθητεία τοπικά πάντα σε τοπικό επίπεδο και έτσι να προπαρασκευάσουμε την περίοδο τη χρονική εκείνη όπου ευελπιστούμε ότι θα σημειωθεί ανάκαμψη και θα πάψει πια η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στις δυναμικές χώρες και πιο δυναμικές περιφέρειες αλλά ευρύτερα. Και κάτι παραπάνω, για παράδειγμα, να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να απασχολούν νέους. Ναι, αληθεύει, μπορούμε να πούμε ότι δύο κυρίως τονίστηκαν πρόσφατα. Μία είναι μια περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο, κατά το ευρωπαϊκό εξάμεινο να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να μεταθέσουν την φορολόγηση από την εργασία αλλά στοχοθετημένα για να ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις είτε για να επιδοτηθούν, να ενισχυθούν οι κοινωνικές εισφορές για τους νέους αν απασχολούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέους στις, ε, στις ε, δραστηριότητές τους ή να υπάρξει ανακούφιση όπως και στην Ιταλία για παράδειγμα αν προσλαμβάνονται νέοι να υπάρχει επιδότηση και βλέπω ότι και για το άλλο και υπήρξαν και κάποιες ε, επιφυλάξεις, το δυναμικό και η δυνατότητα κινητοποίησης Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κύριος Χόγερ, έκανε στεναρές δηλώσεις ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα έχει κύριο ρόλο για στοχοθετημένα δάνεια και πιστώσεις σας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν απασχολήσουν και απασχολούν νέους. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να γίνει και να λειτουργήσει αυτό και η προσπάθεια αυτή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα συνεισφέρει και προς την ευόδοση αυτού του στόχου για την ε, πρόσληψη νέων και να δούμε το δυναμικό που υπάρχει να βελτιωθεί σε σχέση με αυτές τις ενθαρρυντικές ε, δηλώσεις από πλευράς του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τώρα, κάτι άλλο για την παράνομη εργασία Schwarzarbeit Πιθανότατα απάντησα όσο περισσότερο μπορούσα επ' αυτού. Για το green arbeit, πράσινη εργασία. Και αυτή υπάρχει, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, green jobs, πράσινη απασχόληση. <clears throat> Έχει αναγγελθεί στο πακέτο μέτρων, στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, ότι θα πρέπει να εργαστούμε παράλληλα με έναν άξονα προγράμματος δράσης ε, που είχε προαναγγελθεί και τον Απρίλιο ε, πέρυσι, κάναμε περισσότερη πρόοδο για τις ICD jobs, για τις πράσινες ε, θέσεις απασχόλησης. Δημιουργήσαμε ένα μεγάλο συνασπισμό ώστε να προσκληθούν επιχειρήσεις, εταιρείε να συμμετάσχουν σε αυτό το πλαίσιο και να έχουμε και κατάρτιση που θα προετοιμάζει τους πολίτες μας για αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Ωστόσο δεν είναι ένας τομέας μόνο σε όλες αυτές τι δραστηριότητε, αλλά είναι πολυσχηδή τομή δραστηριοτήτων και σύνδεση πολλών τομέων. Αλλά αληθεύει ότι κάποιοι τομείς έχουν περισσότερη ε, εμβέλεια όπως ε, οι οικοδομέ, ε, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τομεί που είναι περισσότερο Έντονη εργασία στο ΜΙΣΕ και θεωρούμε ότι μέσω συνεργασίας του scoreboard των πινάκων επιδόσεων και των δικτών θα μπορέσουμε να έχουμε πρακτικές συγκεκριμένες εξειδικευμένες προτάσεις μέχρι τότε και όταν θα πάω στο Λονδίνο για το σεμινάριο το οποίο η κυρία, Λαμ, η κυρία Λάμπερτ θα προαγάγει, τότε ελπίζω ότι θα είμαι σε θέση να σας δώσω περισσότερα στοιχεία για όλα αυτά, για την προπαρασκευαστική εργασία. Δεν είναι για εφέτος αλλά για του χρόνου που προβλέπετε. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι τότε λοιπόν ώστε να εξειδικευθούν και να αναπτυχθούν αυτά τα αναγκαία στοιχεία και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για αυτά. Να επανέλθω αν έχω ένα λεπτό. Εντάξει, ωραία. Να μπορέσω να, ε, σε ένα μισό λεπτό να απαντήσω για το θέμα των κομμωτών και κομμωτριών σε σχέση με τους κοινωνικούς εταίρους. Λοιπόν, Πολλοί έχουν φύγει, αλλά βλέπω ότι πολλοί άλλοι παραμένουν και ότι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κανένας αυτοματισμός στη διαδικασία και δεν υπάρχει και προθεσμία. Η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει το θέμα, αλλά μια συμφωνία κοινωνικών εταίρων αυτόματα δεν γίνεται ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ούτε, και δεν, ούτε υπάρχει και προθεσμία για να απαντήσει η Κομισιόν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Θα, ούτως ή άλλως η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει διάφορα πράγματα, να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα σε αυτό και στι υπόλοιπε πολιτικές, παραδείγματο χάρη υγεία και ασφάλεια στον χώρο, στο χώρο εργασία, αλλά έξυπνη νομοθεσία και μια διαδικασία refit όπως τη λέμε, επανένταξης του θέματος αυτού δηλαδή, και δεν είναι εύκολο όλα αυτά τα θέματα να τα δούμε και να μην υπάρχουν και συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές. Η Κομισιόν, ε, όπως και το Κοινοβούλιο, ασχολείται με τα θέματα των αρμοδιοτήτων της, δηλαδή ε, της, το κόστος των επιχειρήσεων, την ισο, ισότιμη, ισοτιμία μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, το και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να ικανοποιήσουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ θετικά αυτά τα τελευταία λόγια. Θέλουμε πολύ να συνεχίσουμε αυτόν τον διαθρωμένο διάλογο μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και εξ ονόματος των συναδέλφων που άντεξαν μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς, γυναίκες και άνδρες και την εξαιρετική μας γραμματεία. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας.